Συνάδελφοι, να επανέλθουμε στην συνεδρίασή μας και πριν πάμε στην επόμενη έκθεση της ε, κυρίας ε, Γιάλα Σέντερ, Εδώ πάντα αναζητούμε Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, τους έχουμε λοιπόν από την κάτω Σαξονία ε, μετά την πρόσκληση της κυρίας Μάισνα. Να τους καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή μας. Έχουμε δύο ομάδες. Η πρώτη είναι ήδη παρούσα και η δεύτερη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έρθει αργότερα. Θα ευγνωμονούσα την πρώτη ομάδα να μεταφέρει το μήνυμα του καλωσορίσματος στη δεύτερη ομάδα εμπειρογνωμόνων του συναδέλφους τους και πάλι σας ε, καλωσορίζω σε αυτό το τελευταίο απόγευμα της συνεδρίας της Επιτροπής για αυτή τη φορά. Έχουμε ακόμα κάποια ενδιαφέροντα θέματα στην ημίσια διάταξη. Ελπίζω να βρείτε την συνεδρίαση ενδιαφέρουσα και καρποφόρα. Σε κάθε περίπτωση και πάλι καλωσορίζω την ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Κάτω Σαξονία. Διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ε, η συγγήτρια η κυρία Αγιάλα Σέντε Δεν ήλπιζα ότι θα δούμε τη μέρα που θα το χειριστούμε το θέμα αυτό, αλλά έφτασε η μέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Μπράιαν, πράγματι. Ξανά εδώ, μαζί, καλό αυτό. Το θέμα αυτό το, είχαμε, το είχε εγκαταλείψει το Συμβούλιο, έκθετο, και άλλοι κάποιοι. Να σας υπενθυμίσω, τουλάχιστον ιδιαίτερα σε εσάς που δεν, έχετε, ε, δεν γνωρίζετε τι είχε συμβεί στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού το Μάρτιο του 2011 έκλεισαν τρία χρόνια από τότε που πρώτο παρουσιάστηκε η οδηγία επί Γαλλικής ε, Προεδρίας. Η Γαλλική Προεδρία ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το ζήτημα έτσι ώστε από το Κοινοβούλιο ε, να λήξει η ατιμορρησία των οδηγών οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μια, ε, ε, στη χώρα στην οποία κάνουν παράβαση των κανόνων οδικής ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα έτσι ώστε οι Παραβάσει οι οποίε ε, γίνονται εκτό ε, της ε, χώρας μόνη κατοικία να τιμωρούνται. Υπάρχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε ισχύ ένα σύστημα διμερών συμφωνιών που όμως δεν έχουν δώσει το κατάλληλο αποτέλεσμα δεδομένου ότι η κινητικότητα είναι διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είχε ακολουθήσει μια λογική προσέγγιση, όχι εναρμόνιση ούτε των, των παραβιάσεων, ούτε ε, των αδικημάτων δηλαδή, ούτε των ποινών. Ε, πρότεινε ένα σύστημα ανταλλαγής ε, πληροφοριών που θα επέτρεπε στις αρχές οδικής ασφάλειας να εφαρμόσουν ένα σύστημα που θα οδηγούσε στην τιμωρία και στην επιβολή ποινών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ ευαίσθητο έναντι αυτή της ε, ανάγκη η πρόταση Κομισιόν να ε, βελτιωθεί ε, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη και αυτά τα οποία επιβάλλουν ποινές, ποινικές κυρώσεις όσο και αυτά που επιβάλλουν διοικητικέ κοινώσει παραβιάσει κανόνων ε, οδική ασφάλεια να μπορούν να τιμωρούν τις, τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων. Κατά τη διάρκεια των, του διαλόγου μας ε, προέκυψαν και άλλου τύπου παραβάσει οι οποίε θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν αλλά τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα να διατηρήσουμε τις τέσσερις παραβάσει οι είχε προτείνει η Κομισιόν ε, ταχύτητας, ε, αλκοόλ στο αίμα ζώνες ασφαλείας και παράβαση του κόκκινου σηματοδότη. Αυτές είναι τέσσερις παραβάσεις τις οποίες είχε προτείνει η Κομισιόν και είναι αδικήματα, είναι παραβάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και άλλωστε όλες αυτές μαζί αποτελούν το αντιπροσωπεύουν το 75% των ε, ε, θενατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσουμε να μειωθούν οι θάνατοι ε, στους δρόμους. Στην πρώτη ανάγνωση λοιπόν το Κοινοβούλιο διατήρησε αυτές τις τέσσερις ε, παραβάσεις. Ε, προσπαθήσαμε όμως να συμπληρώσουμε τη διαδικασία, δηλαδή όχι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και τα άλλα απαραίτητα υπόλοιπα βήματα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ε, ποινή θα τιμωρείται. Ότι δεν θα μένει ατιμόρυτος ο οδηγός σε οποιοδήποτε σενάριο. Ε, είτε αυτές οι παραβάσεις επιβεβαιώνονται μέσω ραντάρ είτε μέσω κάμερας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι, γιατί ε, αν συλληφθεί ο οδηγός ε, προφανώς θα πληρώσει το πρόστιμο για να αφαιθεί ελεύθερος. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις που οι ε, παραβάσεις βεβαιώνονται μέσω κάμερας ή ραντάρ. Η ρανταρ ανάγνωση, στην πρώτη ανάγνωση ε, η έκθεση εγκρίθηκε σχεδόν με ομοφωνία, με πολύ πλατιά συνένεση. Διατηρήσαμε τις τέσσερις παραβάσεις, καλύπταμε όλα τα κράτη-μέλη και προτείναμε και μια πλήρη διαδικασία. Ε, με πλήρη προστασία επίσης των ε, προσωπικών δεδομένων. Λάβαμε υπόψη πάρα πολύ το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα Ζητήσαμε την ε, καλύτερη ενημέρωση των οδηγών έτσι ώστε αυτό το σύστημα το οποίο τους ε, επηρεάζει και ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα έτσι μικρό ξεσηκωμό ε, ε να γίνει καλύτερα κατανοητό. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε καλύτερη ενημέρωση των οδηγών. Μετά από την πρώτη ανάγνωση γνωρίζαμε, γιατί μας το είχε πει, μας είχε πληροφορήσει το Συμβούλιο, ότι το Συμβούλιο τα συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη που πάντοτε μας μπλοκάρουν τις πρωτοβουλίες ε, για τη δημιουργία ενός ε, κοινού ευρωπαϊκού χώρου οδικής ασφάλειας άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα. Ε, με ποια δικαιολογία, με ποια αφορμή ότι ε, δεδομένου ότι η οδηγία αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις έδινε λαβή σε ποινικέ διαδικασίες η νομική βάση δεν ήταν αρκετή. Η νομική βάση που είχε προτείνει η Κομισιόν δεν ήταν επαρκής. Μετά μάλιστα και την ε, υιοθέτηση και την έναρξη εφαρμογής της, ε, συνθήκης ε, ε, ε, λέγεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα αστυνομικής συνεργασίας. Καταλάβαμε βέβαια τι υπήρχε πίσω από αυτή την επιχειρηματολογία. αυτό που υπήρχε ήταν ότι το Συμβούλιο είναι αρνητικό σε οποιαδήποτε πρόταση του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εναρμόνιση ε, των ε, παραβάσεων των αδικημάτων και των ποινών ε, καταλάβαμε ότι εκείνη η πρόταση του Κοινοβουλίου δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει παρόλο ότι ήταν πλήρης γιατί ε, κάλυπτε τις ανάγκες όλων των αρχών οδικής ασφάλειας, αστυνομίας, χωροφυλακής κλπ. Το καταλάβαμε ότι δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει, υπήρχε ε, πλειοψηφία, ε, ε, μειοψηφία μάλλον που θα μπορούσε να μπλοκάρει την πρόταση αυτό στο Συμβούλιο ε, και αυτό έγινε σαφές σε, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Προεδρία, πολλές προεδρίες προσπάθησαν να προωθήσουν το θέμα αλλά δεν έγινε κατόρθωτο. Εμείς προσπαθήσαμε να πιέσουμε σε συνεργασία με οργανώσεις θυμάτων κλπ. Δεν άλλαξε όμως η κατάσταση Συμβούλιο μέχρι τον Ιούλιο του περασμένου έτους, του 2010. Η Βελική Προεδρία ε, που είχε φαίνεται αρκετό ελεύθερο χρόνο διότι δεν είχαν προβλήματα με την κυβέρνηση που ήταν απούσα και ανύπαρκτη ε, είχε μια πολύ καλή ευφύ ιδέα Βελική Προεδρία συγκεκριμένα μας ρώτησε αν θα ήταν δυνατόν να ξεμπλοκάρουμε το θέμα μέσω ε, της χρήσης μια διαφορετικής νομικής βάσης. Δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι τότε. Εμείς θεωρούμε ότι η οδική ε, ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνει στην, ε, στο πλαίσιο νομικής βάσης των μεταφορών, αλλά αν δεν αλλάζαμε την νομική βάση, αν δεν βρίσκαμε μια άλλη εναλλακτική λύση, το θέμα αυτό θα έμενε ε, στους αιώνες των αιώνων παρκαρισμένο στο Συμβούλιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να εξετάζουμε αυτή την άλλη εναλλακτική λύση. Ήταν το 2010, μην ξεχνάτε, έπρεπε να αξιολογήσουμε αν είχαμε φτάσει, αν είχαμε πετύχει τον ε, στόχο της ε, μείωσης κατά 50% των θανάτων στους δρόμους ήταν προφανές ότι δεν είχαμε πετύχει το στόχο μας, ε, συνεπώς ήταν επίγον, όλο και πιο επίγον, ε, να υιοθετήσουμε καινούρια να μέσα ε, έτσι ώστε να επιταχύνουμε την βελτίωση της κατάστασης. Συνεπώς ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε, μάλλον είπαμε στο, στην Βελική Προεδρία να ξεκινήσει να σκέφτεται μια, αυτή την άλλη εναλλακτική λύση. Και νομίζω ότι η Βελική Προεδρία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, το πέτυχαν. Κατάφεραν να μετακινήσουν τα εμπόδια. τροποποιώντα την νομική βάση, χρησιμοποιώντα ω νομική βάση την αστυνομική συνεργασία, χωρί βέβαια να ξεχνάμε ότι το πλαίσιο είναι πάντοτε η κοινή πολιτική μεταφορών ή και η κοινωτική πολιτική μεταφορών. Οπότε αυτή ήταν η διέξοδος που βρήκε η Βελική Προεδρία και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κοινή θέση. Βέβαια στο δρόμο, στην πορεία, χάσαμε αρκετά στοιχεία από την αρχική πρόταση. Όμως κερδίσαμε και κάτι. Κερδίσαμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο έκανε ένα πρώτο βήμα. συμφώνησε σε μια πρώτη φάση για την, σύσταση, για την ε, υιοθέτηση ενός τέτοιου κειμένου. Μετά ε, διευρύνθηκε το πεδίο, γιατί αυτά τα τρία χρόνια τα οποία πέρασαν, ευαισθητοποίησαν πολλούς ανθρώπους στο Συμβούλιο. Ε, το θέμα των ναρκωτικών, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που προσθέθηκε. Επίσης, προστέθηκε η μη χρήση κράνους από τους μοτοσυκλωτιστές. Οι μοτοσυκλωτιστές είναι ο τομέας, ας πούμε, η ομάδα στην οποία μικρότερη μείωση έχουμε δει ε, στους θανάτους από τις υπόλοιπες. Ε, επίσης ε, προσθέθηκε το, η παράβαση της ε, παράνομης στάθμης στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και θέματα ασφάλειας αλλά παρεμποδίζει και τη διέλευση άλλων σημαντικών οχημάτων όπως ε, νοσοκομιακά κλπ. Και τέλος προσθέθηκε και η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου. Αυτή η χρήση ε, είναι παράνομη μόνο σε ορισμένα Σε αυτά στα οποία είναι παράνομη ε, θα εφαρμόζεται η οδηγία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που προσθέθηκαν όλα αυτά ε, στο κείμενο που μας έστειλε το Συμβούλιο. Τώρα, φτάνουμε στο αρνητικό κομμάτι. Τι χάσαμε, καταρχήν με την, αλλαγή της νομικής βάσης. Πρώτον, μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η, η νομική βάση αφήνει εκτό τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, που έχουν την ε, δυνατότητα αυτοεξαίρεση. Όταν επήλθε η συμφωνία κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας στο Συμβούλιο, τόσο η Ιρλανδία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι ήθελαν να συμμετάσχουν, να μην αυτοεξαιρεθούν, να συμμετάσχουν και να καλύπτονται από την οδηγία. Εδώ μεταξύ είναι μια συζήτηση και εσείς κύριε Σίμψον την ξέρετε πολύ καλύτερα και ακούστηκαν πολλές ε, φωνές ε, αντίρρησης και η κυβέρνηση δεν κατάφερε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κατάφερε ε, να εντάξει τη χώρα στην κάλυψη αυτής της οδηγίας. Η Ιρλανδία από την άλλη μεριά και εκεί η πολιτική κατάσταση δεν τους επέτρεψε να συμμετάσχουν παρόλο ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Σε ό,τι αφορά τη Δανία προς το παρόν τα πράγματα είναι σε εκκρεμότητα. Ελπίζουμε ότι μέσω διμερών συμφωνιών να εφαρμοστεί το σύστημα και στη Δανία. Αυτή είναι η πρώτη σημαντική αδυναμία του νέου συστήματος. Η δεύτερη αδυναμία έχει σχέση με το ίδιο το σύστημα. Η συνολική διαδικασία που είχαμε προβλέψει εμείς στην πρώτη ανάγνωση, δηλαδή ανταλλαγή, από την ανταλλαγή των πληροφοριών μέχρι την ε, υιοθέτηση των ποινών στα πλαίσια βέβαια πάντοτε της επικουρικότητας, το είχαμε προβλέψει και αυτό. Όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η αλυσίδα δεν εγκρίθηκε, οπότε το Συμβούλιο παρέμεινε στην ανταλλαγή πληροφοριών και μόνο. Αυτή είναι η μόνη υποχρέωση. Τώρα από εκεί και πέρα το κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει τη διαδικασία όπως το επιθυμεί. Το Συμβούλιο δεν αποφάσισε τίποτα επί αυτού του ζητήματος. Το Κοινοβούλιο είχε προβλέψει όλη τη διαδικασία, αλλά το Συμβούλιο ε, την ε, περιόρισε στο πρώτο βήμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Τώρα, τι πρόταση κάνω εγώ. Ε, καταρχήν είμαι αισιόδοξη. Έτσι, είμαι αισιόδοξη γιατί αν δεν ήμουν αισιόδοξη δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Τώρα, σταθμίζοντας τα συν και τα πλήν, τα υπέρ και τα κατά. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξανά έναν στόχο για τη μείωση των ε, θανατηφόρων ατυχημάτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Επίσης έχουμε προσθέσει το στόχο της μείωσης των τραυματιών. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας καινούρια μέσα και εργαλεία. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο ε, ακόμα και για αυτό το πρώτο βήμα το οποίο δημιουργεί ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμεύσει έτσι ώστε να δημιουργεί μια δυναμική συνεργασία ανάμεσα στις αρχές οδικής ασφάλειας. Κάτι τέτοιο ε, θα μας υποσχόταν πολλά για το μέλλον ενδεχομένως να ε, παρατείνουμε και να διευρύνουμε αυτό το σύστημα. Οπότε ως εισηγήτρια ε, επιθυμώ να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι θα παραπλανούσαμε τους πολίτες αν τους λέγαμε ότι αυτό το οποίο έθεσε το τραπέζι μας το Συμβούλιο είναι χρήσιμο για την επίτευξη του στόχου της εξάλληψης ατιμορρησίας. Αυτό που μας προτείνει το Συμβούλιο έχει μια κέρια δυναμία. Αν το κράτος μέλος το οποίο λαμβάνει τις πληροφορίες δεν θελήσει να δώσει συνέχεια, τίποτα δεν μπορεί να του το απαγορεύσει. Οπότε, αυτό που έχουμε κάνει είναι, μέσω των τροπολογιών μας, ε, να προσθέσουμε μια ε, ρήτρα ε, αναθεώρησης για την συνέχιση του συστήματος. σε συνεργασία με την ε, Κομισιόν. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές, για παράδειγμα τις οδηγίες χρόνου εργασίας, μέσω, της, ε, μέσω των οποίων κατευθυντήριων γραμμών ε, ενισχύεται η εφαρμογή της. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. Επίσης με την τροπολογία που προτείνουμε η ε, η πληροφόρηση να γίνεται όχι μόνο προς την Κομισιόν αλλά και προς τα κράτη-μέλη. Ε, επίσης, έχω υποβάλει και μία ακόμα τροπολογία ε, που, είναι, που έχει σχέση με το εξή. Η ογκρική Προεδρία έχει, έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας, τεχνική ομάδα εργασίας και ένα σύστημα, το σύστημα εύχαρης, το οποίο ζητούμε να ε, προσαρμοστεί στις ανάγκες της οδικής ασφάλειας. Το παράδειγμα 1 1α έχει το καλό ότι αν εφαρμοστεί θα ανακτήσουμε τις ε, χώρες που... Ζητώ συγγνώμη πρόεδρε μακρηγορώ, αλλά ε, πρέπει να ενημερώσω τους συναδέλφους που δεν ήταν ευρωβουλευτέ στην προηγούμενη θητεία μα. Με αυτό το σύστημα του παρατήματο 1 1α ε, έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τον Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Ακόμα και χωρίς να γίνει ένα επίσημο opt-in. Οπότε είναι πολύ καλή η δουλειά της Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, ήταν πολύ καλή κυκλονομιά που πήρε από το Βέλιο βέβαια. Επίση ζητάμε την ενίσχυση προστασίας των δεδομένων, παρόλο ότι το ε, ισχυρό σύστημα είναι αρκετά ισχυρό. Νομίζω είναι σημαντικό να το ε, ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτά νομίζω. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσει, με χαρά θα σας ακούσω. I thank you. No, no, that's why I was quite happy to let you go <laughs> for for a while. Ναι, ξέρω ότι έχουμε παρακολουθήσει το θέμα τρία χρόνια τώρα και περιμέναμε από το Συμβούλιο κάποιες ε, αντιδράσεις ε, και πράγματι τα νέα μέλη καλό είναι να πληροφορηθούν τα όσα είχαμε περάσει στην προηγούμενη φάση. Επομένως έχετε δίκιο. Τώρα οι σκιώδεις ε, εισηγητές θα μιλήσουν. Καταρχάς ο κύριος Μπάχα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, δεν είμαι και τόσο νέο μέλος της Επιτροπής. Ε, έχω βέβαια κληρονομήσει αυτό το θέμα και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα Σέντερ, να τη συγχαρώ, ο ιδίως για την επιμονή της, διότι να ασχολείται κανείς τρία χρόνια με ένα θέμα, όντως απαιτεί πολύ ισχυρή δύναμη και ουσιαστικά εδώ ε, έχουμε να κάνουμε δύο διαφορετικές πολιτικές. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα είναι πολύ πιο φιλόδοξο και θέλει να το προωθήσει και όντως κάπου να καταλήξει σχετικά με την οδική ασφάλεια και ε, δεν θέλω εδώ να πω ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να βελτιώσει την ε, οδική ασφάλεια αλλά είναι πιο ρεαλιστές και δέχονται μόνο αυτά που είναι ε, εύκολα εφικτά. Και φαντάζομαι ότι σαν ε, Επιτροπή δεν πρέπει αυτό να μας ε, αποθαρρύνει διότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να ακολουθήσουν την ίδια οδό με μας και ε, γι' αυτό βρήκαν την αλλαγή της νομικής βάσης για να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών αλλά αυτό χωρίς να σημάνει ότι θα επιβληθούν και ποινές. Το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε και πιστεύω ότι σαν Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουμε να ε, εφαρμόζουμε αυτή τη φιλόδοξη πολιτική. Όσον αφορά τα ε, διάφορα σημεία όπου έχουμε διαφορές, νομίζω ότι όσον αφορά την νομική βάση δεν έχουμε πρόβλημα ε, αν περάσουμε από το άρθρο 71 στο άρθρο 87 ε, για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τα νομικά συστήματα των χωρών. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό γιατί αντιλαμβάνουμε ότι διαφορετικά δεν θα μας ακολουθήσει το Συμβούλιο Χωρί χωρίς να ξεχνάμε όμως ότι μετά από λίγο καιρό θα διαπιστώσουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα ε, ε, μεταφορών σχετικά με την οδική ασφάλεια και να μην το ξεχνάμε και να θυμόμαστε ότι ε, κάλλιο αργά παρά ποτέ να καταλήξουμε σε μία τροπή η οποία να μας ικανοποιεί. Όσον αφορά την ρήτρα επεξεργασίας ε, εμείς λέμε 6 μήνες, το Συμβούλιο λέει 36 μήνες, αλλά κατά τις διαπραγματεύσεις ελπίζω ότι θα υπάρξει μία προσέγγιση, πρέπει να βρεθεί μία προσέγγιση, διότι το άρθρο αυτό 25 δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε, πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι, κατά τρόπον ώστε να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για συγκεκριμένες εκθέσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά με το άρθρο 28 αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τις διαπραγματεύσεις διότι το Συμβούλιο Βεβαίω, δεν θέλει να το αναγνωρίσει όπως εμείς θα θέλαμε. Δεν έχουν δηλαδή προβλήματα μόνο με τους υπουργούς ε, ε, δικαιοσύνης αλλά και μεταφορών και εσωτερικών στις διάφορες χώρες για να υπάρξει η εφαρμογή και κατά τις ε, διαπραγματεύσεις πιστεύω ότι η τύχη είναι με το μέρος μας και ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση πρέπει να επιμείνουμε θα κάνουμε ε, όσον αφορά το συνολικό σύστημα, ε, πιστεύω ότι το σύστημα των ανταλλαγών πληροφοριών δεν έχει καταρτιστεί κατά τρόπον ώστε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα συσσωρευτούν να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι θέλουμε να υπάρξει ένα ε, λογισμικό, μία επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμη και εάν στην ε, πρώτη φάση η ανταλλαγή πληροφοριών είναι δωρεάν και απλή. Ε, όσον αφορά τα άλλα θέματα θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ ιδιοκτήτων του ε, οχήματος και των οδηγών διότι για τη σχέση αυτή υπάρχουν διαφορές αναλόγως των ε, χωρών και πρέπει να δούμε εάν ε, εμείς θα είμαστε υπέρ του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του οδηγού. Ε, μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι τρεις χώρες οι οποίες διαφωνούν θα ακολουθήσουν ε, την ε, οδό για να συνεργαστούμε στο θέμα της οδικής ασφάλειας γιατί δεν θα θελήσουν να μείνουν αποκλεισμένες επί του θέματος αυτού πρέπει να κοιτάξουμε να μειώσουμε τον αριθμό των νεκρών και πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών, νομίζω ότι μπορούμε να χαιρετήσουμε την πορεία που διαγράφεται. Σήμερα το πρωί για τα ναρκωτικά αναγνωρίζουμε Είσαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και οι αριθμοί οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί μας έπεισαν ότι είναι τρομακτικοί και επ' αυτού συμφωνούμε με το Συμβούλιο ότι αυτή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής πρέπει να ισχύσει. Φαντάζομαι τώρα ότι κατόπιν αυτού μπορούμε να εκφράσουμε την πλήρη εμπιστοσύνη μας και στήριξη στην εισηγήτρια και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σαβισάρ, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Πολύ ευχαριστώ που μετά από τόσοι οι οποίοι περνάμε στη δεύτερη ανάγνωση, να, σας, ξεκινήσω όμως ε, εξηγώντας σας γιατί η Επιτροπή Μεταφορών χρειαζόταν αυτή την οδηγία. Γιατί χρειάζεται να αυξήσουμε την ασφάλεια και να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα. Συνεπώς, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ε, να διαθέτουμε κυρώσεις και οι κυρώσεις να εφαρμόζονται. Δεν είναι αρκετό να επιβεβαιώνουμε τις παραβάσεις αλλά να μην επιβάλλουμε κυρώσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επιτευχθούν και τα δύο. Εγώ είμαι προφανώς ε, πιο φιλόδοξη γιατί είμαι νέο μέλος και γι' αυτό το λόγο νιώθω πιο απογοητευμένη από τη συγγήτρια. Λυπούμε που η, η συγγήτρια συμφωνεί ε, με, το Συμβούλιο να αλλάξουμε την νομική βάση. Νομίζω ότι πολύ εύκολα υποχωρούμε και δεχόμαστε αυτή την ε, και δεχόμαστε ότι το ζήτημα εμπίπτει στην αστυνομική συνεργασία. Δεν νομίζω ότι το Κύπρο θα μας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων μας. Στην τροπολογία 25 βέβαια η συγκήτρια αναθέτει στην Κομισιόν ε, τα επόμενα τρία χρόνια να συλλέγει και να, στοιχεία και να αναλύει με τα τρία, τρία χρόνια μετά δηλαδή την υιοθέτηση της, ε, της οδηγίας ε, να αναλύει στοιχεία για το κατά πόσο θα είναι απαραίτητη η αλλαγή της νομικής βάσης αλλά αυτό δεν είναι αρκετό Ε, επίσης προτείνει, προτείνεται ε, ανταλλαγή στοιχείων μέσω του εύχαρης. Ε, ίσως αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαδικασίες, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και αυτό στο κείμενο. Επίση θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τα 19, 20 και 21, να τροποποιήσουμε τα 19, 21 που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Αυτή τη στιγμή είναι αντιφατικά. Θα έπρεπε να τα ξαναδούμε. Επίσης δεν δέχομαι την πρόταση του παρατήματο 1 1α. δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, αρκετές πληροφορίες. Θα ήταν αρκετή απλώς η ενημέρωση από πλευράς των αστυνομικών αρχών ότι το συγκεκριμένο άτομο διέπρεξε τη, μια συγκεκριμένη παράβαση, τίποτα παραπάνω. Ως φιλελεύθερη, πιστεύω ότι θα έπρεπε να δίδεται μεγαλύτερη ε, να, να εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ε, ελευθερία του ατόμου και είναι ε, θα πρέπει να αποφεύγουμε υπερβολικές, ε, τη συλλογή υπερβολικά πολλών πληροφοριών. Εφόσον οι διαδικασίες δεν έχουν ξεκινήσει, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο άτομο διέπραξε μια συγκεκριμένη παράβαση. Νομίζω ότι ε, προ... προέχει το κριτήριο το τεκμήριο της αθωότητας. Εφόσον ακόμα κανείς δεν έχει, ένας κάποιος δεν έχει καταδικαστεί, δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να πάμε πιο μακριά από το κείμενο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, καταρχήν αυτή η οδηγία απέβλεπε ε, να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε ποινές διασυνοριακά και να υπάρξει κάποια πειθαρχία μεταξύ των οδηγών. Αυτή ήταν ε, η αιτία που μας ε, οδήγησε να θελήσουμε να βελτιώσουμε τα θέματα ασφαλείας της οδήγησης. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επιμονή με την οποία προσπάθησε να προωθήσει το θέμα αυτό και σχετικά με την αντίσταση την οποία αντιμετωπίζουμε ε, από το Συμβούλιο έχω πλήρη κατανόηση διότι τώρα έχουμε φτάσει και επιτύχει μία βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. Ε, και τι θα γίνει παρακάτω. Δηλαδή, ε, κάποιος ο, αυτός ε, πηγαίνει με 180 χιλιόμετρα στην χώρα που κάνει διακοπές ενώ όλοι οι άλλοι πάνε σαν τις χελώνες με 100 δεν τιμωρείται αλλά κινδυνεύουν και οι άλλοι πράγμα που δεν ενδιαφέρει το Συμβούλιο και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στάση του Συμβουλίου δηλαδή κάθε προσπάθεια καταστέλλεται, καταστρέφεται και δεν συμφωνώ καθόλου εάν συνεχίσουμε έτσι δεν έχει πλέον κανένα νόημα να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών όταν ούτως ή άλλως τα πάντα το Συμβούλιο τα απορρίπτει και δεν προχωράμε. Όσον αφορά την αλλαγή της νομικής βάσεως και θα ήθελα να επανέλθω και εδώ. Δεν είναι το πιο βασικό θέμα, είναι όμως ένα σύμβολο του τι συμβαίνει διότι εδώ μιλάμε απλώς για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκτελεστικών δυνάμεων και τίποτα παραπάνω. Όλα τα άλλα θέματα της ασφαλείας των συγκοινωνιών δεν συζητούνται διότι δεν μιλάμε πλέον για, για αύξηση της ασφαλείας αλλά απλώς για ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, πολύ αρέσει στο Συμβούλιο να κάνει τέτοια πράγματα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι απαιτεί η ανταλλαγή πληροφοριών. Και πάντοτε υπάρχει μία σαφής απόρριψη από, πολλά, από πολλές χώρες. Πολλές χώρες που έχουν πολλούς τουρίστες ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν μας δίνουν τα εργαλεία κατά τρόπον ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όσον αφορά τις μεταφορές, δυστυχώς ο καθένας πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός στην Ιφίλιο και οι άλλοι κάνουν όλοι τα λάθη. Ε, όταν ρωτάει κανείς κάποιον θα σας πω ότι το 80% θεωρούν ότι είναι καλή οδηγία ενώ δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Κανείς δεν παραδέχεται τα λάθη του. Ε, και στα κράτη-μέλη το ίδιο συμβαίνει. Το κάθε κράτος πιστεύει ότι εφήβρε την πυρίτιδα και ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι ή ανίδεοι και δεν τα καταφέρουν τόσο καλά ώστε ο κάθε στη χώρα του. Μπορούμε να κάνουμε ατελείωτες εκστρατείες πληροφόρησης αλλά δεν θα πετύχουμε τίποτα εάν ε, δεν ε, μπορέσουμε να επιβάλλουμε τις απαιτήσει μας και να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία ζητούμε. Υπάρχει και ένα άλλο βασικό θέμα. Μέχρι στιγμής για τα περισσότερα ναρκωτικά δεν υπάρχει υπάρχει ε, κανένα ανεγνωρισμένο ενιαίο ε, μέσον ε, για να δοκιμάσει κανείς εάν υπάρχει χρήση ναρκωτικών. Και δεν ξέρω αν φταίνε τα κράτη-μέλη ή όχι, αλλά ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση είναι τα φάρμακα. Ορισμένα φάρμακα δεν λαμβάνονται οικειοθελώς και δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις τους και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακόμη επαρκώς επιλύσει. Ε, γενικώ νομίζω ότι στα γενικά θέματα κυκλοφορίας σωστό είναι να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να έχουμε μία ενιαία νομική βάση. Αλλά αν δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος επιβολής κυρώσεων δεν πάμε πουθενά. Και βλέπουμε τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να βελτιώσουν την κυκλοφορία με το να υπάρχει διασυνοριακά ένα ένας ενιαίος τρόπος επιβολής κυρώσεων. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να το διακηρύξουμε για να καταλάβουν ε, οι πολίτες ότι δεν ευθύνονται όλα τα θεσμικά όργανα της Ενώσεως αλλά σαφώς και απαρεμβάτως μόνο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ινές για την ποιότητα εργασίας της και την αντοχή της και να της πω αμέσως ότι συμφωνώ με τον μηχανισμό που προτείνει αλλά έχω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, ως αυτά το μηχανισμό αυτομάτου ελέγχου μπορούμε να διατυπώσουμε και να, και να γράψουμε το αυτοκίνητο το οποίο ευθύνεται προβλέπεται για την ε, παράβαση αλλά όχι τον οδηγό και αυτό είναι ε, περίπλοκο. Αυτό υπάρχει στη Γαλλία και στη Γαλλία λένε ότι εάν δεν υπάρχει καταγγελία θα ε, τιμωρήσουμε τον οδηγούς και αυτό είναι πολύ λεπτό σε ευρωπαϊκή κλίματα και θα είναι ενιαίο για όλους τους αυτόματους ε, μηχανισμούς. Το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε το, την επίστολη πολύ πληροφόρησης που έχει προσωπικά ευπαθή στοιχεία. Δηλαδή η γυναίκα μου μπορεί να ανοίξει μία επιστολή και να δει ότι με γράψανε στο Παρίσι τη στιγμή που υποτίθεται ότι ήμουν στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν ένας χαρακτήρας εμπιστευτικών πληροφοριών και θα πρέπει, βέβαια θα μου πείτε ότι έπρεπε να, μείνω, να κάτσω στα αυγά μου και να μην ξενοκοιτάω. Αλλά ε, η γυναίκα μου ουσιαστικά ε, είχε, ε, ήταν αυτή που γράψανε στο Παρίσι και εγώ νόμιζα ότι ήταν στις Μετά, όσον αφορά τα δεδομένα, ξέρετε ότι ε, ε, υπάρχει τρόπος ε, να περιλάβετε τα στοιχεία σε μία τράπεζα δεδομένων μπορείτε να τους τσακώσετε σε κάποια διόδια. Πόσο καιρό όμως θα μπορεί ο καθένας να κρατήσει αυτά τα δεδομένα, παραδείγματο χάρη τις πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν διότι μπορεί να τιμωρηθούν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν, πώς θα μεταφέρουμε τα δεδομένα και πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούμε τα δεδομένα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι πολύ ανησυχητικά. Η κυρία Μάισνερ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην περίπτωση αυτή ε, έχουμε να κάνουμε με ένα φάκελο τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ο ένας χαίρεται ε, ε, αν τη γλιτώσει και τη σκαπουλάδι δεν το γράψουν δηλαδή και από την άλλη πλευρά μιλούμε για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, πώς μπορούμε να μειώσουμε τα ατυχήματα της κυκλοφορίας και να μην έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα στο δικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε διάφορα θέματα σε διάφορες χώρες και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ δεν τα βρήκε εύκολα, το ξέρουμε, γιατί ε, βάσει της επικορικότητας έχουμε αρμοδιότητες για την ε, νομοθεσία και τη ρύθμιση και για το θέμα το δικό πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εναρμονίσουμε και να συγκρίσουμε. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι στο καλό δρόμο, δεν θα γιατί έχουν ήδη λεχθεί πολλά. Πρέπει να δούμε εάν ε, πάμε σωστά ή πρέπει να δούμε πού μπορεί να αποτύχουμε στο Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ εγώ υποχρεωτικό να συμβεί, αλλά στο 1β υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, για τους ελέγχους του ινοπνεύματος ή την υποψία ε, ε, ελέγχους σε περίπτωση υποψίας κατανάλωσης ινοπνεύματος Μόνο εάν ε, συντονίσουμε τις προσπάθειες σαν κράτη θα μπορούμε να ε, επιτύχουμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνονται σωστά οι ανταλλογές στοιχείο βεβαίως προστατεύοντας τα στοιχεία, αλλά αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει και στην Ευρωπόλ και αλλού. Ε, πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα και είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ να συγχαρώ την κυρία Αγγέλα Σέντερς για την ε, έκθεσή της. Εμείς την περιμέναμε την έκθεση αυτή και περιμέναμε και την εφαρμογή της οδηγίας εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια κάποιων προεδριών στο Συμβούλιο δεν ανελήφθησαν βήματα στο φάκελο αυτό, υπήρξε δισταγμός. Τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας ε, δημιουργεί μια νέα νομική βάση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο φάκελο αυτό γιατί πιστεύω ότι η οδική ασφάλεια θα, θα έπρεπε να είναι μέρος του, του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να ασκήσουμε την όποια επιρροή μπορούμε στις κυβερνήσεις μας για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή γιατί θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις θα πρέπει να σεβαστούμε το θέμα της οδικής ασφάλειας και σε διασυνοριακό επίπεδο. Χρειάζονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης, χρειάζονται ευφυή συστήματα μεταφορών και προφανώς προσπαθούμε να μην αφήσουμε εκτός καμία λεπτομέρεια που να αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά στο επίπεδο που διατηρούνται τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, ως εισηγήτρια και για το θέμα του κανονισμού πρόσβασης στις οδικές μεταφορές, είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται στους οδηγούς. Ο κανονισμός όμως αυτός δεν επιβάλλει μόνο ποινές και κυρώσεις στους οδηγούς, αλλά και στις επιχειρήσεις των οποίων οι οδηγοί κατ' εξακολούθηση παραβιάζουν τους ε, κανόνες οδικής ε, κυκλοφορίας. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να εκφράσω την υποστήριξή μου στην έκθεση της κυρία Αγιάλα Σέντερ και ίσως να τα πετύχουμε. Η κυρία Φώστερ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Εγώ δεν ε, ομιλώ εξ ονόματος της ομάδας, αλλά σε μια οπτική βρετανική αν θέλετε. Εμείς αποφασίσαμε να μην ε, συμμετάσχουμε αν θέλετε. Ε, θυμάμαι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε λάβει η χώρα, γιατί προερχόμαστε από τελείως διαφορετικές νομικές βάσεις και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα εδώ. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι θα αλλάξουμε όλη την ε, δικαστική, αν θέλετε, διαδικασία σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Και για παράδειγμα, μιλώντας για το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι ότι δεν τονίζουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας, είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό. Ορισμένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν, οι τυχαίοι έλεγχοι κτλ. σίγουρα έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο η νομική δυσκολία που επισέρχεται είναι ότι μπορούμε να ασκήσουμε δίωξη μόνο κατά του οδηγού, όχι του ιδιοκτήτη του οχήματος. Έτσι έχουν τα πράγματα νομικώς μιλώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σχετικά με την ποσοτικοποίηση της επιβολής της κύρωσης αν θέλετε. Αν υπάρχει δηλαδή χρηματική κύρωση ή τι άλλο είχαμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι το σύστημα με τους βαθμούς, το point system, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο συμμόρφωσης, για να το πούμε έτσι. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της, των αρμοδιοτήτων των αστυνομικών αρχών. Είναι και η αστυνομία και η τροχέα δηλαδή τι κάνει σχετικά με το θέμα σε σχέση με την όποια κύρωση ή δίωξη του οδηγού ή του ιδιοκτήτη του οχήματος. Και αναφέρομαι εδώ και στα προσωπικά δεδομένα που λέγαμε πριν, γιατί είχαμε και σχετικά ε, περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δεν διώκουμε τον ιδιοκτήτη σε κάθε περίπτωση, αλλά μόνο τον οδηγό. Εμείς οπωσδήποτε έχουμε δεσμευτεί να συμμετάσχουμε σε μια προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας αλλά στο μεσοδιάστημα αυτή είναι η κατάσταση που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπωσδήποτε σημειώνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ο κύριος Κράμερ, δύο λεπτά. Λοιπόν, υπάρχει μια κατάσταση ότι υπάρχουν Γερμανοί που ζουν στο Λονδίνο και στη Στοχόλμη και πηγαίνουν στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητό τους γιατί κανείς δεν θα τους πιάσει. Και αυτό δεν είναι σωστό και επίσης πρέπει να είναι αναγκαία η προστασία των στοιχείων και ε, όπου υπάρχει πολιτική υπάρχει και ο σωστός δρόμος να ε, προστατεύσουμε τα δεδομένα διότι ε, μπορέσαμε να συνανοηθούμε με τους υπεύθυνους συγκεντρώσεις δεδομένων για το χρόνο που θα αποθηκεύει κανείς τα στοιχεία αυτά. Το τελευταίο όμως θέμα που θίξατε, δηλαδή αν είσαστε είμαστε με το αυτοκίνητο σε μια άλλη ε, ε, ε, πόλη και σας γράψουν για υπέρβαση ταχύτατος. Στην Γερμανία όμως κάποιος καταψήφισε αυτήν την διάταξη και δεν έχει διαμορφωμένη γνώμη από αυτούς. Διότι ένας ένας ε, ο οποίος κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είναι παράνομα ε, σταθμευμένο θα πληρώσει το πρόστιμο αν τον πιάσουν και μετά θα τον πληρώσει ο οδηγός που άφησε το αυτοκίνητο και βγήκε έξω. Λοιπόν, ε, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες μεταφοράς της ευθύνης και γιατί πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ των σταθμευμένων αυτοκινήτων από αυτών που κυκλοφορούν δεν το καταλαβαίνω, χρειάζεται όμως πειθαρχία. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για οδική ασφάλεια και έχουμε και εδώ και πάλι μία χωρισμένη Ευρώπη. Μιλάμε για Ενωμένη Ευρώπη, για Single European Sky και δεν τα βρίσκουμε για την ξηρά. Εγώ για δύο λεπτά. Εγώ συμφωνώ με τον Λιχτεμπέργκερ με την ε, κυρία Λίχτεμπεργκερ, συγγνώμη. Ε, περιμέναμε τρία χρόνια για το Συμβούλιο και ε, είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν αφορά την νομική βάση. Ε, δεν έχει σχέση με το κατά πόσον διώκουμε το αυτοκίνητο τον οδηγό. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αυτό είναι το ζήτημα. Στο ενωμενο Βασίλειο η κόρη μου ε, την κόρη μου την έπιασε ε, μια κάμερα για ταχύτητα ε, και το πρόστιμο ήρθε σε μένα, γιατί εγώ είμαι ιδιοκτήτης και, τι, και εγώ πήγα και τους είπα, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο, είναι η κόρη μου και τελικά ε, χρεώθηκε στην ίδια. Συνεπώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, ψευτινές δικαιολογίες ε, αυτά της κυβέρνησής μας. 70.000 ε, μη Βρετανοί πολίτε διαπράττουν αδικήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια κάθε χρόνο στην Ηνωμένο Βασίλειο και δεν διώκονται. 70.000, 71.000 συγκεκριμένα. Και έχουμε την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι θα τιμωρούνται, όπως τιμωρούνται από το Βρετανικό νόμο, όλοι οι Βρετανοί πολίτες. Και τι κάνει η κυβέρνησή μας, αυτό εξαιρείται. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουμε επιτόπου πληρωμή των προστήμων, όμως οι Βρετανοί υπήκοοι ε, μπορούν να υποχρεωθούν να πληρώσουν επιτόπου τα πρόστιμά τους όταν οδηγούν σε άλλες χώρες. Οπότε η αυτοεξαίρεση είναι ε, διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Βρετανών, με κάτι τέτοιο. Συνεπώς το θέμα δεν είναι νομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πιο συγκεκριμένα έλλειψης πολιτικής βούλησης. Τώρα, ένα σχόλιο για τα όσα είπε η κυρία Σάβησα για την αλλαγή της νομικής βάσης. Φαίνεται σαν να υποχωρούμε προς την, πολιτική, προς την αστυνομική συνεργασία ε, με την αλλαγή της νομικής βάσης. Αλλά υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Ο λόγος είναι ότι ήμασταν σε αδιέξοδο με την αρχική νομική βάση. Ε, μα μακάρι να άλλαζαν από μόνα τους τα πράγματα, αλλά προτιμώ το 1% από κάτι παρά το 0% ή το 100% του τίποτα. Συνεπώς είναι θέμα συμβιβασμού. Ε, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μία θέση, μια κοινή θέση, χρησιμοποιώντας την αστυνομική συνεργασία, αυτή την καλή ιδέα της ε, Βελικής Προεδρίας. Αλλά βλέπετε ακόμα και έτσι και με αυτές τις αλλαγές εξακολουθούμε να έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να αυτοεξαιρεθούν. Οπότε η συγκήτρια είναι σωστή. Παρόλο που καταλαβαίνω και τα άλλα επιχείρηματα. Το, το πιο ισχυρό όμως επιχείρημα υπέρ του κειμένου είναι ότι μιλάω με τους αστυνομικούς διευθυντές ε, στην Ευρώπη και βλέπω ότι το θέλουν. Θέλουν μια τέτοια νομοθεσία. Ε, ακόμα και αυτοί που είχαμε ε, στο πρωινό, ο Μάικλ θα το επιβεβαιώσει, είχαμε κάποιους αστυνομικούς διευθυντές το πρωί στο πρωινό και μας το είπαν και αυτοί. Ε, θέλουν να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα. Όπως είπε και η κυρία Γιάλα, μην περιμένουμε όμω το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί εκεί είναι θέμα πολιτικών επιλογών. δεν θα μαλώσουμε. Είπε εσύ τα δικά σου, είπα και εγώ τα δικά μου. Κομισιόν. Thank you, Mr. President. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε αυτό το δύσκολο φάκελο του τελευταίους μήνες και ειλικρινά ελπίζει και εύχεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα τα ενδιαφερόμενα με συγχωρείτε μέρη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να επιτεθεί μια συμφωνία. Εκτιμούμε πραγματικά τις προσπάθειες της εισηγήτριάς σας ε, για να γίνει μια θετική συνεισφορά για τον Ευρωπαίο πολίτη στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Στους άτυπους τριλόγους ε, που θα γίνουν και γίνονται, πάντα είναι διαθέσιμη η Κομισιόν και έτοιμη να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Αλλά πολύ συνοπτικά να σας πω την ε, θέση μας σχετικά με τις ε, τροπολογίες. Για το τεχνικό παράρτημα 1α, η τροπολογία 27, θεωρούμε ότι η τροπολογία αυτή καθιστά προστιθέμενη αξία απέναντι στην πρόταση του Κοινοβουλίου. Είχε γίνει λόγος και για την 17 και 18, ιδιαίτερα 18, που διευκρινίζει τα θέματα τα σχετικά με την επιστολή πληροφόρησης. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ε, αρχής επανεξέτασης έτσι όπως προτείνεται και στην τροπολογία 25, αλλά πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι διατηρούμε υπόψη ε, το δικαίωμα πρωτοβουλίας βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα, τις πτυχές προστασίας δεδομένων ε, είμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης της διατάξεως αλλά να προειδοποιήσω κατά της νομικής ασάφειας, της έλλειψης ασφάλειας δικαίου δηλαδή, και των υφισταμένων νομοθεσιών σχετικά με το θέμα. Εμείς σημειώνουμε ε, τα του άρθρου 4 ε, με την επιφύλαξη της ε, νομικής εξέτασης του κειμένου και είμαστε επίσης υπέρ των τροπολογιών για τις αιτιολογικές σκέψεις. Για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αισιόδοξη ότι η προσέγγιση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ είναι μια πολύ καλή βάση για να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση και η οδηγία αυτή όταν εγκριθεί θα διευκολύνει πραγματικά την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του ε, κώδικα κυκλοφορίας. Γνωρίζετε την σημασία που εμείς θεωρούμε ότι έχει το θέμα και ότι έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για να ελεγχθεί ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων και θανατηφόρων ατυχημάτων πάνω απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχετε υπόψη σας και την ε, προετοιμασία της ε, Λευκής ε, Βίβλου με το υπογραμμιζόμενο όραμα το, της Zero Vision δηλαδή την κατακόρυφη μείωση και έλεγχο των ατύχηματων. Εμείς προσβλέπουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει κάτι να προσθέσει σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο να ευχαριστήσω απλώς τους ε, συναδέλφους ε, που τοποθετήθηκαν σε αυτήν την μακρά δικασία. Είναι αλήθεια ότι είχαμε αρχικά βάση την, δώσει την ε, νομική βάση ως θετικό σημείο κίνησης για το Συμβούλιο αλλά να διαβεβαιώσω και την κυρία Σάρ και του υπόλοιπου συναδέλφου ότι για την τροπολογία 25 δεν είχαμε ποτέ ξεχάσει το ζήτημα και νομίζω, νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση. Πράγματι υπάρχει διάκριση του ιδιοκτήτη και του οδηγού αλλά έστω και με κάποιες επιφυλάξεις είχε επιληθεί εν μέρη το ζήτημα και το έντυπο που θα ε, μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και το οποίο είναι το πιο εύχριστο, αν θέλει, το πιο πρακτικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διευκολύνει τα πράγματα, νομίζω ότι εν μέρει επιλύει, εν μέρη επιλύει την κατάσταση, αν και είναι αλήθεια ότι υπάρχει το θέμα, το πρόβλημα της προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων, υπάρχει το σύστημα ε, αλλά έτσι, ως τέτοιο μάλλον, δεν υφίσταται, θα πρέπει ε, να τροποποιηθεί για τις συγκεκριμένες παραβάσεις τις οδικές. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος να εφαρμοστεί αυτούσια. Ωστόσο, είναι ένα σύστημα που έχει δικλείδες ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και το ενισχύουμε, είμαι βεβαίως ανοιχτή, σε οποιαδήποτε άλλη τροπολογία μπορεί να το ενισχύσει υπεραιτέρω. εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή αντίφαση. Προς τον κύριο Ρικέ να πω ότι είμαστε σύμφωνοι με τα σχόλια αυτά, αλλά και υπό την ε, δική σας ε, προεδρία όπου είχαμε ξεκινήσει με αυτό το νομικό κείμενο, ήταν πράγματι η Γαλλική Προεδρία που πραγματικά κατέβαλε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να προωθήσει το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά την ε, ανταλλαγή δεδομένων υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν φόρμουλες για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε γρήγορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το εξακριβώσουμε και θα το επαναξετάσουμε. Και να πω επίσης στον κύριο Σίμψον ότι είναι αλήθεια και δεν είναι θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά αν είχαμε και κάποιον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, για το επόμενο ένος εγώ θα είμαι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά και ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε εκείνα τα εκρεμή ζητήματα που τρία χρόνια τώρα παραμένουν εκρεμή. Έτσι για να κλείσουμε μια θετική νότα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, προθεσμία είναι η 18η Απριλίου με την ψήφο για τον Μάιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Το επόμενο σημείο στην μέση διάταξη λοιπόν, <laughs> εξίσου δύσκολο και αντιφατικό, ο κύριος Ντεγκράντες και η έκθεση του επί την ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών με ειδική εμφάση στους ερωτές σώματος. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή έχουν υποβληθεί 190 τροπολογίες από 30 συναδέλφους. Κάτι που αποδεικνύει την σημασία της έκθεσης αυτής, του θέματος αυτού. Το θέμα έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο και πολύ συζητημένο. Θα προσπαθήσω να αποφύγω της ε, σύγκρουσης. Ευχαριστώ πολύ που ε, αφιερώσατε χρόνο και θα αφιερώσω και εγώ χρόνο στην ανάλυση και στην... θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλα τα όσα προτείνετε. Είναι πολλές οι τροπολογίες, ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Πιστεύω ότι είμαι πεπισμένος ότι συμπίπτουμε σε πάρα πολλά πράγματα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι αδύνατον να δούμε λεπτομέρως όλες τις τροπολογίες αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά θα χάσουμε όλο μας το απόγευμα. Νομίζω το πιο χρήσιμο θα ήταν να μην μπω σε λεπτομερή ανάλυση. Θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο να αξιολογήσουμε σε ομάδες, σε δέσμες τις τροπολογίες και επί αυτών να τοποθετηθούμε. Επί των, και κυρίως επί των θεμάτων των πιο αφιλεγόμενων προκύπτων. Σαρωτές. Λοιπόν, κάποιοι μέσω τροπολογιών θέλουν να μην εγκατασταθούν σαρωτές σώματος. Μέσω τροπολογιών ε, επιχειρηματολογούν με τον ΑΒ β τρόπο για να δικαιολογήσουν τη στάση τους. Να πω το εξή. Ότι σέβομαι τη γνώμη τους, αλλά δεν τη συμμερίζομαι. Συνεπώς, ως εισηγητής θα τοποθεθώ εναντίον τέτοιων τροπολογιών. Αν βέβαια είναι επικοδομητικέ και βελτιώνουν την έκθεση, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν θέλουν να αποτελούν δικαιολογία. Ξεκινώ από την εξή θέση. Οι σαρωτέ αποτελούν προστιθέμενη αξία στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες μας. Δεύτερον, ε, λέγεται ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το δικαίωμα στην προσωπική ζωή και με τη χρήση τους δεν θα πρέπει να βλάπτουν την υγεία, τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν θα πρέπει να καταστρέφονται αμέσως χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης. Το θέμα είναι τα χαρακτηριστικά των σαρωτών. Πρέπει να είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα η χρήση να είναι αναλογική έναντι του κινδύνου που ε, σκοπεύουμε να, από τον οποίο σκοπεύουμε να προστατευτούμε. Αυτά είναι οι στόχοι μας. Ε, συμβαστικά, τι μπορούμε να προτείνουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, σε, μεγάλα, σε μεγάλες δέσμες τροπολογιών οι οποίες μοιάζουν μεταξύ τους. Πρώτον, ποια τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείτε θεωρώ ότι δεν πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά μιας οποιασδήποτε τεχνολογία με την οποία πειραματιζόμαστε στην Ευρώπη εκτός. Γιατί αυτό θα ήταν η υπέρβαση καθήκοντος. Υπάρχει όμως μια γενική συνένεση μέσω από όλε τι τροπολογίες και αυτή είναι να αποκλειστεί η χρήση των ακτίνων Χ. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά τον ακτίνων χ, αλλά τελικά οι απόψει συμφωνούν. Οπότε προτείνω μια συμβαστική φόρμουλα, έτσι ώστε να αναφέρουμε στο Συμβούλιο πως πρέπει να αποκλειστεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας. Δεν είπα να απαγορευτεί. Δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει απαγόρευση της χρήσης μιας ε, ε τεχνολογίας γιατί θα ξεφεύγαμε από το κοινοτικό δίκτυο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, απεικόνηση του ανθρωπίνου σώματος. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε απεικόνηση η οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της ε, ε, ασφάλειας. Θα ήθελα να αποφύγουμε οποιαδήποτε αναφορά στην ανθρώπινη σιλουέτα. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι μια ανησυχία η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί. Ε, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών, ε, ε, δεδομένων. Ναι, ασφαλώς, πάντοτε υπάρχει, υπάρχουν τέτοιου είδους ανησυχίες. Οι τροπολογίες συμφωνούν με τη δική μου θέση. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να συσσωρεύουν τα, τα δεδομένα ούτε και να αποθηκεύονται. Εδώ δεν υπάρχει συμβασμό. Δεν θα πρέπει να γίνεται αποθήκευση. Όχι να γίνεται αλλά να περιοριστεί η χρήση τους. Όχι. Να χρησιμοποιούνται επί τόπου και να μην αποθηκεύονται πουθενά. Τίποτα άλλο. Εκεί δεν υπάρχει θέμα συμβασμού. Αυτό θα ζητήσουμε. Τεχνολογικά θέλουμε να μην γίνεται καμία αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ε, σαρωτές οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα συσσόρευση εικόνων, ε, διατήρησής τους δηλαδή ή αποθήκευσής τους. Έτσι κι αλλιώς πάντως εμείς θα ζητήσουμε να μην γίνεται κανός είδους διατήρηση ή αποθήκευση. Μετά, υγρά. Μεγάλο θέμα. Όπως γνωρίζετε, πάντοτε έλεγα για τα υγρά ότι το, όχι για τα γενικά, ότι το, το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι λογικό στις απαιτήσει του και στα αιτήματά του. Αλλά θέλω να κάνω την εξή διάκριση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μια πρώτη ημερομηνία, 29 Απριλίου, και μετά η ημερομηνία του 2013. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, στο εξή, στο θέμα του 2013. Ειλικρινά όμως να σας πω ότι για, για τον α ή τον β λόγο που δεν θα κρίνω, πολλές χώρες δεν θέλουν ε, να υλοποιηθεί, να τεθεί σε ισχύ η 29η Απριλίου, αυτή η ημερομηνία. Η Κομισιόν θα πρέπει να πάρει, να αναλάβει τις ευθύνες της όμως. Εμείς θέλω να επαναλάβουμε την προσήλωσή μας για το πώς πρέπει να είναι το 2013 ε, ε, η κατάσταση. Τώρα, να μαλώσουμε εμείς για το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί με το Duty Free 29 Απριλίου, δεν, δεν είναι εκεί το θέμα. Ε, θα, κατά την άποψή μου είναι άχρηστη αυτή η και θα μπορούσε και να διαγραφεί κιόλα. Γιατί η, έτσι κι αλλιώ η γνωμοδότηση θα εγκριθεί μετά τι 29 Απριλίου. Ε, Α αναλάβει τι ευθύνε τη η Κομισιόν, όπω όπως πρέπει, όπως αρμόζει. Γιατί να μπούμε σε μια σύγκρουση στην οποία συγκρούνται συμφέροντα τα οποία είναι άσχετα με εμά. Τώρα, και πέρα. Για το 2013 μπορούμε να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό εκεί πέρα. Ε, μη διάκριση. Υπάρχει μια βασική συμφωνία. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πιο πολλές συμφωνίες παρά διαφωνίες. Ε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το α ή το β επίθετο, την α ή τη β διατύπωση, αλλά η ουσία είναι ίδια. Θα μπορούσαμε να ε, ξεκαθαρίσουμε το θέμα της μη διάκρισης με ένα συμβασμό. Οι συμβασμοί βέβαια θα πρέπει να διατυπώνονται εις τρόπον ώστε να αισθάνονται ικανοποιημένοι όλοι όσοι έχουν ζητήσει τροποποίησης. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ρητά να αναφέρουμε ότι δεν θα γίνεται κανένας είδους διάκριση γιατί υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν πως μέσω με διάφορα παραθυράκια οι ρογμές μπορούν ε, να ε, ε, γίνουν παραβάσεις αυτού του κανόνα με διακρίσει με βάση το φιλετικό προφίλ ή οτιδήποτε άλλο. στην ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας υπάρχει η έννοια του υπόπτου, αλλά εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το πράγμα. Ε, εμείς δεν πρόκειται ε, να ασχοληθούμε με την αντιτρομοκρατική δράση. Γιατί μια τρομοκρατική δράση έτσι κι αλλιώς δεν αποκαλύπτεται, έτσι. Γιατί αν μόλις την αποκαλύψει πάβει να είναι τρομοκρατική δράση. Συνεπώς εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το θέμα. Ε, βάρος. Απόδειξης και αλληλογραφία. Ε, το θέμα αυτό δεν μπήκε στην έκθεση ε, χωρίς λόγο. Προέκυψε διότι στην αρχή μιλούσαμε για σαρωτές, ε, ενώ μετά αρχίσαμε να μιλάμε και για υγρά και για βάρη και για, ε, και για ναύλους, ε, για ναύλους και για αεροπλάνα μεταφοράς αλληλογραφίας. Δηλαδή διευρύναμε το πεδίο εφαρμογής μας. Οπότε ε, χρειάστηκε να ζητήσουμε από τους τεχνικούς να μας πούν τι μπορεί να βελτιωθεί, τι μπορεί να γίνει ε, και σε αυτούς τους τομείς. Αρκότερα θα δούμε ε, και άλλα θέματα με τις παρεμβάσεις σας, αλλά να σας πω ε, και κάτι άλλο. Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλοι συμφωνούμε. Αλλά ορισμένοι ε, από τους συναδέλφους τοποθετούν αυτό το θέμα σε διάφορες τροπολογίες. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα μόνο σε ένα σημείο του κειμένου. Δεν είναι δυνατόν να είναι ρεφρέν αυτό. Γιατί αλλιώς η έκθεση θα γίνει δυσανάγνωστη. Θα μιλήσω με όλους όσους ε, απασχολεί το θέμα αυτό, ε, έτσι ώστε να βρούμε μια συμβαστική λύση, έτσι ώστε αυτοί που ανησυχούν να ε, ικανοποιηθούν και θα δεχτώ το θέμα των μελλοντών δικαιωμάτων να μπει στην έκθεση. Δεν, δεν είναι καθόλου προβληματικό. Τώρα, σαρωτές σώματος, σαρωτές προστασίας. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ το αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό το ζήτημα. Εγώ ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη χρήση της α ή της β ορολογίας. Ε, το 2008 μιλούσαμε για σαρωτές σώματος, μετά η τεχνολογία άλλαξε και τώρα μιλούμε για σαρωτές προστασίας. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ακριβής ο όρος πλέον. Αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Τώρα εσεί θέλετε να επιστρέψουμε στου σαρωτές σώματο. Δεν συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Να σα πω την αλήθεια, εμένα το ίδιο μου κάνει. Απλά ο όρο που χρησιμοποιείται από του τεχνικού, από του εμπειρογνώμονε, είναι σαρωτέ προστασία. Εφόσον έχουμε ε, μια συμφωνία του επιστημονικού κόσμου για αυτό το ζήτημα, ε, πρέπει και εμεί να την ακολουθήσουμε. Σέβομαι την άποψή σα, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι σωστέ οι τροπολογίε αυτέ που έχετε υποβάλει. Έχετε υποβάλει πολλέ τροπολογίε το θέμα αυτό κάποιες από τις τροπολογίες σας θα τις υπερψηφίσω έτσι, αλλά κάμε κάποιες άλλες διαφωνώ. Δύο πραγματάκια μένουν ακόμα και τελειώνω, πραγματικά ειλικρινά πρόεδρε. Πληροφόρηση, εκ των προτέρων πληροφόρηση ε, του επιβάτη. Το αναφέρει η έκθεση, το παραλαμβάνουν πολλοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό. Ο επιβάτης που θα περάσει από σαρωτή θα πρέπει να γνωρίζει αναλυτικά ποια είναι τα δικαιώματά του. Το λέμε. Και αν κάποιος συνάλφο χρειάζεται κάτι παραπάνω, συμβιβαστικά να, το, να βρούμε μια λύση. Συμφωνούμε σε αυτό. Μετά, κατάρτιση προσωπικού, το ίδιο. Είναι θέμα κλειδί. Στις νέες τεχνολογίες πάντοτε είναι σημαντικό να, να παρέχουμε κατάρτιση στο προσωπικό τόσο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού, όσο και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τον επιβάτη που βλέπει ορισμένα του δικαιώματα να υποσκάπτονται μερικές φορές. Τέλος, προτείνουμε στην γραμματεία στις 9 Μαΐου, αν είναι δυνατόν και συμφωνείτε, να, κάνουμε μια συνάντηση έτσι ώστε να συζητήσουμε τις συμβεστικές προτάσεις. 9 Μαΐου λοιπόν ή ε, οποιαδήποτε άλλη στιγμή ε, πιο κατάλληλη βρει η γραμματεία. Ακόμα και αν υπάρξουν ε, τροπολογίες οι οποίες δεν θα συμπεριλάβω στις συμβαστικές προτάσεις, θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους οι οποίοι τις έχουν υποβάλει, έτσι ώστε να ε, μιλήσω μαζί τους προσωπικά και να τους εξηγήσω τη στάση μου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεγκράντης. Να πάω στους σκιώδεις ηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Φλέκενστάιν. Θα δώσω στους σκιώδεις εισηγητές τέσσερα λεπτά στον καθένα και θα δούμε για τους υπόλοιπους, γιατί προστίθενται συνέχεια ομιλητές στον κατάλογο. Κύριε Φλέκενστάιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω δεν χρειάζομαι καν τα τέσσερα λεφτά, διότι στην πολιτική ομάδα δεν υπάρχει ακόμη αποκρισταλωμένη γνώμη. Ε, με παρεκάλεσαν οι ε, με παρεκάλεσε ο σκιώδης εισηγητής ο κύριος Λάιχτφρικ να, πει, να πω λίγα λόγια γιατί είναι στην Αυστρία σήμερα. Ε, έχει υποβάλει 11 <clears throat> τροπολογίες τις οποίες ε, ως επτοπλίστων έχει προσυπογράψει με άλλους συναδέλφους και πρέπει να τις χωρίσω σε κατηγορίες ε, για να ε, τις κατατάξω όπως το έκανε και ο κύριος Δεγκράντες. Καταρχήν ο κύριος Λάιχτφριντ δεν θα ήθελε να υπάρξει καταγραφή των στοιχείων η η χρήση των ε, ε, ε, ακτίνων πρέπει να αποκλειστεί και είναι αστείο οι άνθρωποι να σκανάρονται είναι κάτι το οποίο να αντιμετωπίσετε με μεγάλη χαλαρότητα αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς του τους ανθρώπους όπως την αλλογραφία ή τα εμπορεύματα και επίσης όσον αφορά την νομοθεσία που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την ε, το σχέδιο μάλλον, ε, το νομοσχέδιο σχετικά με την ε, αποζημίωση για την ε, αεροπορική ασφάλεια γιατί θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό το υπερψηφίσαμε. Εγώ κατάγομαι από το Αμβούργο. Δύο φορέ την εβδομάδα λοιπόν έχω τη χαρά να βλέπω έναν body scanner. Ε, μία φορά λειτουργεί, μια δεν λειτουργεί. Ε, δεν λειτουργεί το πρωί γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιβάτες ε, την ώρα που φεύγω νωρί και κλείνουν το μηχάνημα γιατί είμαστε πολλοί και την νύχτα όταν γυρίζω περνάμε από το σκάνερ Οπότε ε, ε, στη συνέχεια το 90% ψηλαφούνται επιπλέον. Οπότε όσον αφορά τις ε, τροπολογίες 28 και 29 έχω μεγάλη συμπάθεια όπως άλλως και η τροπολογία 171. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια στα αεροδρόμια και για τους ανθρώπους και για τα εμπορεύματα που συνδυάζονται με τους ανθρώπους και ε, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα body scanners, στους ανιχνευτές του ανθρωπίνου σώματος. Διότι πιστεύω ότι ίσως μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς από ό,τι θα θέλαμε, διότι αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμή στα αεροδρόμια δεν αρκεί για να μας κάνει να αισθανθούμε ασφαλείς και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι όμως πολύ απλό να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Σίμψον, δηλαδή ότι το σκάνερ είναι απλώς ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε στην εργαλειοθήκη μας και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε διότι στη συνέχεια ε, υπάρχουν ορισμένοι που συνδυάζονται με ακτίνες Ράντκεν ε, όπως δηλαδή η ακτινογραφία και πρέπει αυτό να μείνει στη διάκριση των κρατών μελών και να δούμε πώς θα γίνει. Αλλά αν θέλει κανείς ε, ε, να ανοιχνεύσει πράγματα μέσα στο σώμα με ακτινογραφία θα χρειαζόταν τόση ακτινοβολία ώστε θα ήταν απαράδεκτη γι' αυτό και προς στιγμής ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικέ λύσεις που θέλουν ακόμη να συζητηθούν. Αυτό που θα ήθελα εγώ ήταν ότι δεν χρειάζεται να σαρώσει κανείς ολόκληρο το σώμα. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε και αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο εξαιρετικά και δεν θέλουμε να καταγράφονται επιπλέον όλα αυτά τα στοιχεία Επ' αυτού έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες και λέμε ακριβώς αυτό. Αλλά στην Γερμανία, στο Λουμπέκ, πήγα στην αστυνομία και εξετάσαμε επί τρεις ώρες τι γίνεται για να δούμε ότι δεν υπάρχει βλάβη για την υγεία του ανθρώπου και αν προστατευόμαστε ως προς τα στοιχεία. Βεβαίως καλό είναι να ελέγξουμε και άλλες τεχνικές ε, για το πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ε, ε, κρικτικά. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για το 34. Η κυρία Φώστερ μίλησε για το profiling, αλλά ό,τι έχει σχέση με τα στοιχεία, όπως και με τα στοιχεία για το, τα, αεροπορικά ταξίδια που εξετάζει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, πρέπει να δούμε πώς συνάδουν με την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων διότι μας λέγουν ότι στο Αμβούργο αργεί να εγκατασταθεί το σύστημα το ξέρω πήγα και εγώ εκεί ε, και αν δεν είναι όριμο ένα σύστημα δεν μπορεί να ισχύσει, πρέπει να το βελτιώσουμε και θα θέλαμε να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Για το τροπολογία 93 νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ακόμη και ε, εκτός σε ειδικέ περιπτώσεις που πρέπει να προστατεύονται για εγγύους, για παιδιά κτλ. Διαφορετικά πρέπει να δούμε αν αν δέχεται κανείς να περάσει από τις ακτίνες ή θέλει να υπάρχει άλλος, άλλο είδος εξετάσεως με ψηλάφιση κτλ συζήτηση σαν μικροφόνου. Αν έχουμε υποψίε ούτω ή άλλω ε, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε για να τον εξετάσουμε και να ε, μπορούμε να έχουμε τα pictograms. Ε, δεν πρέπει όμως επουδενή λόγο να υπάρξει εικόνα ολοκλήρου του σώματο και όπως σα είπα γενικά δεν θα θέλαμε την αποθήκευση των στοιχείων και με την τροπολογία 45 θα ήθελα να πω ότι αν υπάρξει μια εικόνα πρέπει κανείς να τη συνδέσει ε, άμεσα με τον ενδιαφερόμενο και όχι να την αποθηκεύσει. Και επίσης ε, αυτό που είπαν ορισμένοι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των σκάνερ και τέλος για τα εμπορεύματα ε, είπα ότι καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε την οδηγία 300 του 2008 των ταχύτερων δυνατών γιατί στα φορτία πολλά δεν γίνονται που θα έπρεπε να γίνονται και ε, αν έχουμε αποφασίσει κάτι και ε, έχει υπερψηφιστεί πρέπει και να εφαρμόζεται. Κυρία Λίχτενβέργκερ. ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκτενή παρουσίαση της ε, γνωμοδοτήσεώς του. Για μένα Υπάρχει ένα ουσιαστικό επιχείρημα. Εδώ έχουμε μία νέα ονομασία. Δεν ονομάζεται πλέον body scanner γιατί αυτό περιγράφει αυτό το οποίο γνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη αλλά τώρα λέγεται προσωρινά σκάνερ ασφαλείας. Λες και ήταν κάτι καινούριο. Οπότε αυτό που είναι γνωστό από, την, ε, ε, ε, από το 1984 από τη βιβλιογραφία το να βγάζει κανείς ένα νέο όνομα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι καινούριο και δεν είναι υποχρεωτικό να το δεχτούμε. Πρόκειται για ένα body scanner και όχι για ένα σαφή ε, σκάνερ. Γι' αυτό και εγώ έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες απλώς για να αλλάξουμε το όνομα. Εφόσον πρόκειται για body scanner πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μετά για τις ακτίνες Röntgen. Συμφωνώ με όλους αυτούς οι οποίοι είπαν και το τόνισε σαφώς και η Επιτροπή Ελευθεριών ότι η χρήση των ε, ακτίνων Röntgen αποκλείεται για εξετάσεις ρουτίνας γιατί έχει επιπτώσεις επί της υγείας και γι' αυτό πρέπει να λέμε όχι ευχαριστώ, φτάνει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα για εξετάσεις ρουτίνας διότι διαφορετικά θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας και όσο πιο συχνά ταξιδεύει κανείς τόσο περισσότερο κινδυνεύει όσο χαμηλή και να είναι η δόση των ακτίνων Ρόγκεν γιατί βλέπουμε ότι η πραγματική τιμή είναι πολύ ψηλότερη από αυτή η οποία δηλώνεται. Άρα εγώ αποκλείω τελείω τι ακτίνες ρόντκεν. Μετά, προστασία των στοιχείων και αυτό πρέπει να υφίσταται πλήρως και ελπίζω θα μπορέσουμε να πούμε σαφώς ότι δεν θα υπάρξει μια διατήρηση των στοιχείων αυτών, δεν θα συσσωρεύονται τα στοιχεία αυτά, διότι ε, τότε προχωράμε προς το profiling όπου θα συγκεντρώνουμε και άλλα στοιχεία, να δούμε ε, τι βιβλία διαβάζει ο καθένας και όλα αυτά να τα συνδυάζουμε για να διαμορφώσουμε ένα προφίλ κάποιου. Ε, αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι το θέμα του προσωπικού που πρέπει να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας, να έχει καλύτερη εκπαίδευση γιατί σε αυτήν την οδηγία ground handling ε, γίνεται, ε, μία προστακά, ε, γίνεται ένας προς τα κάτω ανταγωνισμός δηλαδή όλο και πιο επαχθείς αμοιβέ σε συνθήκες εργασίας και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ασφάλεια. Άρα επ' αυτού θα πρέπει να επέμβουμε είναι πολύ σημαντικό και αυτό το ξέραμε και από τα τελωνία. Ποιος ανεκάλυπτε κάτι, αυτοί που είχαν πείρα και που είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση και την πείρα για να ανοιχνεύουν. Όσον αφορά την ε, πολιτική ασφαλεία στις αεροπορικές μεταφορές από πλευράς ε, κόστους και από πλευράς ε, εκπαιδεύσεως του προσωπικού πρέπει να εξεταστεί πολύ πιο επιστημονικά. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά τα θέματα αυτά κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην βιβλιοθήκη, στο μουσείο όπου παρουσιάζεται η Μόνα Λίζα και άρα Άρα πρέπει κανείς να σκέπτεται και λίγο παραπέρα στις άλλες εκδοχές και ε, γι' αυτό θέλω να στηρίξω τους συναδέλφους στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ε, ευρωβουλευτές που είναι πολύ πιο προσεκτικοί και εγώ θα ήθελα να σας πω να αναρωτηθούμε δεν υπάρχουν άλλες τεχνικές που να είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές χωρίς να επεμβαίνουν στα προσωπικά δεδομένα και δεν ε, δυσχεραίνουν την κατάσταση περισσότερο διότι εάν ξέρουμε τα πάντα περί ενός ατόμου πρέπει να δούμε τουλάχιστον τι γίνεται ή στα αεροπλάνα και τι ακολουθεί έναν επιβάτη όταν μπαίνει μέσα στο αεροσκάφος. Σας ευχαριστώ λίγο ο Πρόεδρος, και κυρία Φώστα για τους ε, συντηρητικούς. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι έχουν δίκαιο ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή. Υπάρχει ευρεία συνένεση από αυτού και το βλέπουμε διατρέχοντας τις ε, τροπολογίες σε ό,τι αφορά το που βρισκόμαστε. Ο Πέτερ Βαντάλεν είναι επισήμως ο σκιώδης συγητής και μάλλον υποστηρίζουμε οι τροπολογίες ο ένας του άλλου αλλά σε σχέση με τον αριθμό των τροπολογιών είμαστε αρκετά περιορισμένοι Υπήρξα η συγγέντρια και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και προσπάθησα να διατηρήσω μια κάποια συνέπεια μεταξύ των δύο. <clears throat> Αλλά για το αντικείμενο. Πράγματι, έχει δίκαιο η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Είναι σε ρωτή Και εφόσον είναι, ας τον αποκαλέσουμε έτσι. Και είναι ένα πρόσθετο εργαλείο στη θέσή μας για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Τελεία. Πώς λοιπόν το χρησιμοποιούμε καλύτερα. Αυτό είναι το αντικείμενό μας. Είναι σωστό να θέτουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και θα επαναλάβω απλώς ε, τα αρχικά μου σχόλια που υπάρχουν και σε διαφορετική τροπολογία εδώ, ότι πρέπει να τονιστεί το θέμα της συλλογή δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο πληροφοριών μάλλον και όχι δεδομένων και ακόμα παρότι κάποιοι συνάδελφοι δεν συμφωνούν των ε, πληροφοριών profiling ταξιδευτών, ταξιδιωτών. Γιατί όσο περισσότερα στοιχεία θα έχουμε, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την τεχνολογία. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τα θέματα της υγείας. Όλοι έχουν την απόψή τους. Γνωρίζουμε ότι έχουν, υπάρχουν τεχνολογίες ε, στη διάθεσή μας που δεν θα γύρουν ζητήματα ε, προστασίας της υγείας, αλλά σε σχέση με την απεικόνηση ο μόνος, λόγος, ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η απεικόνηση, αν κάποιος χρειάζεται να ε, ε, κρατηθεί για παράδειγμα, Αλλά από τη στιγμή που θα διαγραφεί μια εικόνα ε, μόλις εξέλθει το, το άτομο από το σαρωτή, τότε δεν υπάρχει θέμα αποθήκευση στοιχείων. Τώρα για την ακτινοβολία. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, έγγραφο από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια για την ε, διάχυση εκτινοβολίας σε σχέση με την ε, τεχνολογία των συστημάτων αυτών και πρέπει να το διατηρούμε υπόψη. Γεγονό είναι ότι αν έχουμε εξοπλισμό στη θέσή μα, ο οποίο να μην είναι αντιφατικό στη χρησιμοποίησή του, τότε δεν χρειαζόμαστε να βλέπουμε και εξαιρέσει. Πρέπει να έχουμε τεχνολογία στη θέσή μα που να μην μα υποχρεώνει να έχουμε ομάδες εξαιρέσεων. Ότι δεν πρέπει να περνούν από τους σαρωτές για διάφορους λόγους. Ποιος είναι ο λόγος του να έχουμε ένα σαρωτή σώματο εάν η μισή δεν μπορεί να περάσει για λόγους υγείας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία κάνουμε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους. Και υπάρχει τεχνολογία, το ξαναλέω. Και δύο ακόμα λεπτομέρειες θα έλεγα πρέπει να φτάσουμε σε μια απόφαση σχετικά με το αν αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή όχι. Γιατί το όλο νόημα στην συζήτηση εδώ είναι αν, κράτος, αν κάποιο κράτος μέλος μας πει όχι, είναι προαιρετικό και προτιμούμε να μην το εφαρμόσουμε σε σχέση με ένα άλλο κράτος μέλος όπως το δικό μας, το οποίο αποφάσισε εδώ και καιρό να το εφαρμόσει, αν έχουμε δηλαδή μεγάλο αριθμό επιβατών που δεν διέρχεται από του ερωτέ, τότε τι νόημα έχει η συζήτηση. Είτε έχουμε ένα εργαλείο στη θέσή μα κατά πολέμηση τη τρομοκρατία, προηγμένο τεχνολογικά, χωρί να είναι οχληρό, χωρί να είναι κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, τότε δεν έχει νόημα. Ή μάλλον δεν υπάρχει κίνδυνο του να συζητούμε για το ποιοι θα περνούν. Ή είναι πρόβλημα για την υγεία ή δεν είναι. Εάν χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία που δεν είναι πρόβλημα, τότε μπορούμε να έχουμε του ανθρώπου όπω μα είπε ο συνάδελφο ότι α, όχι, προτιμώ να μην περάσω, προτιμώ να μου κάνουν έλεγχο μέσω ψηλαφίσεω. Το νόημα εδώ είναι ότι να εξεύρωμε τι λύσει που θα μα επιτρέψουν να χρησιμοποιούμε τεχνικά μέσα που να παρακάμπτουμε την, την αναγκαστική ψηλάφιση, να μην τη χρειαζόμαστε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση της προαιρετικότητας ναι εμεί το θέλουμε, άλλοι δεν το θέλουν. Γιατί αλλιώ πραγματικά δεν έχει νόημα η όλη συζήτηση, ούτε έχει νόημα η Επιτροπή να κάνει το οτιδήποτε. Είτε είναι απαραίτητο αυτό το μέσο, είτε α το αφήσουμε. Και συμπερασματικά πρόεδρε και κλείνω, νομίζω ότι έχουμε μια ευρεία συνένεση εδώ, απλώ να σκεφτούμε πιο προσεκτικά πώ θα προχωρήσουμε προ τα εμπρό. Ευχαριστώ η κυρία Βίλς. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο, ο, ο εισηγητής, ε, ε, οι σαρωτές αυτές αντί για body scanners θα έπρεπε να λέγονται ε, security scanners, δηλαδή ασφαλείας. Ε, Αν ναι, πρόκειται όμως να ονομαστούν σαρωτές ασφαλείας θα πρέπει να αλλάξουν όνομα. Έχουν όμως μεγαλύτερη ασφάλεια διότι μπορούν να σαρώσουν τις βασικές σωματικές επιφάνειες και όχι το εσωτερικό. Η τροπολογία 73 της κυρίας Αγίας Αγιάλα Σέντερ επίσης πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί οι, ε, οι σαρωτές αυτές και ο κύριος Φλέκενστάιν πολύ σωστά μας έθεσε το παράδειγμα του Αμβούργου και εγώ είμαι από το Αμβούργο και το έχω ζήσει το ε, σκηνικό αυτό. και βλέπουμε σε ορισμένα αεροδρόμια που έχουν κλείσει τους, ε, τα μηχανήματα αυτά. Επίσης ε, λέγεται ότι δεν πρέπει να βλάπτουν την ε, υγεία τα μηχανήματα αυτά αλλά δεν είναι φιλικά προς την υγεία εν πάση περιπτώσει και αυτό δεν οφείλεται στην έκθεση η οποία καταρτίζεται διότι υπάρχουν ακτίνες οι οποίες επιβάλλονται επιβαρύνουν το ανθρώπινο σώμα και βλάπτουν την υγεία εάν οι ακτινοβολίες αυτές συσσωρευτούν. Ε, συμφωνούν πολύ ότι οι εικόνες αυτές δεν πρέπει να αποθηκεύονται. Είδαμε όμως ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένη διότι όπως όλα τα συστήματα υπολογιστών μπορεί κανείς να τα παραποιήσει και ορισμένοι να έχουν πρόσβαση. Είναι τελείως ε, ανεδαφικό ότι θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια. Επίσης ε, όσοι, όσοι επιβάτες δεν δέχονται να περάσουν από τον σκάνερ ε, δεν είναι σωστό να μην μπορούν να επιβιβαστούν του αεροπλάνου. Ποτέ δεν θα είναι τόσο ασφαλή η έλεγχης η η έλεγχη ε, Μία λύση θα ήταν ίσως να μην ε, πετάει κανείς, αλλά θα πρέπει ε, να υποκείμεθα μόνο σε υπεύθυνε διαδικασίες και έχω υποβάλει 22 τροπολογίες στα θέματα τα οποία έθιξα. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι το θέμα όντως δεν είναι εύκολο και κατά τη γνώμη μου το αντιμετώπισε με κάποια απόσταση και πολύ αντικειμενικά. Για να επανέλθουμε στην αρχή, ε, όλοι γνωρίζουμε περί τύρος όρεκειται, αλλά ορισμένα θέματα τα ξεχνάμε, ε, διότι ε, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει τους ελέγχους, μετά είχαμε το θέμα των body scanner και μετά ε, ξεκίνησε η εξέταση των ε, εμπορευμάτων. Η πολιτικοί λοιπόν ε, αντιδρούσαν εκ των υστέρων, άπαξε κάτι απεκαλύφθη. Πιστεύω λοιπόν ότι με την έκθεση αυτή δεν δίνουμε την εντύπωση ότι αύριο θα είναι οι αεροπορικές ε, συγκοινωνίες ασφαλείς. Πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες και καταρχήν να τις κοιτάξουμε υποκειμενικά, να μην ξεχνούμε την επικορικότητα, διότι κάθε ε, κράτος θα μπορεί αύριο το πρωί να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας και εδώ είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιδράσει στην κατάσταση εάν κάποιο κράτος ε, δεν εφαρμόσει τις αποφάσεις που θα ψηφιστούν τώρα. Διότι αν δούμε ότι μόνο ένα ή δύο κράτη πρόκειται να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, το δεν αξίζει να κάνουμε τόση συζήτηση και αν η κατάσταση διαφέρει τόσο πολύ από τη μια χώρα στην άλλη και υπάρχει καυγάς, δεν νομίζω ότι είναι σε μας ε, το θέμα να το συζητήσουμε εάν πρόκειται όλοι να το απορρίψουν στη συνέχεια. Επίσης όσον αφορά την υγεία Πιστεύω ότι κανείς δεν περιμένει ότι αύριο το πρωί θα ξέρουμε αν είναι βλαβερό για την υγεία του καθενός. Για μένα υπάρχουν ερωτηματικά και πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ελέγχου και σε ορισμένες περιπτώσεις ο επιβάτης έχει ε, το δικαίωμα να αρνηθεί να υποβληθεί σε ορισμένους τεχνικούς ελέγχους και θα έχει δίκιο πιστεύω ότι όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη πρέπει να την παρακολουθούμε. Διότι όπου ε, προχωρήσαμε είδαμε ότι αυτά που μας λέγουν δεν είναι πάντοτε σωστά και η πραγματικότητα προτρέχει. Ας μην ε, προσπαθούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε ορισμένες μεθόδους θα πρέπει πάντοτε να μπορούμε να προσαρμοστούμε και να εξασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν τρία λεφτά αυτά κύριε Γκρός, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ο κύριος Μπράντμπαρν τώρα. Καταρχήν να πω ότι θα πρέπει να οπισθοδρομήσουμε λίγο. Να πάμε λίγο στο παρούμε γιατί μιλάμε. Πριν από λίγο χρόνια είχαμε τους κοινούς κανόνες ε, στη, για την ασφάλεια της αεροπλοείας ε, και ε, οι επιβάτες ε, είχαν δικαίωμα να περιμένουν θα εξασφαλίζεται η ίδια ασφάλεια σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο, από οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πετούσαν. Ε, τώρα, έτσι όπως το γίνεται η κατάσταση, βλέπω ότι δεν θα έχουν τους ίδιους κανόνες. Ε, α, για παράδειγμα, εδώ με τους ε, σαρωτές σώματος. Συμφωνώ με την κυρία Ρίχτεμπεργκερ καταρχήν. Πρόκειται για σαρωτές σώματος. Ας τους αποκαλούμε όπως είναι το όνομά τους, αυτό που είναι. από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σημαντική συνένεση σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να γίνει. Να σας πω για δύο-τρία πράγματα την άποψή μου όμως. Ε, κάποιοι μίλησαν για τη τεχνολογία των ακτινών κλπ. Ας ε, καταρρύψουμε ένα μύθο. δεν είναι το ίδιο να περνά από ένα σαρωτή με το να δέχεσαι ακτινοβολία για 5 λεπτά σε ένα αεροπλάνο όταν πετά. Όχι, δεν πρόκειται για την ίδια ακτινοβολία. Άλλη ακτινοβολία ε, περνάει από το σώμα σου όταν περνά από ένα σαρωτή και άλλη ακτινοβολία που υπάρχει στο περιβάλλον σου όταν πετά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επικίνδυνο μύθο και είναι ε, και η ε, τεχνολογία αυτή έχει ε, σημαντικό, μπορεί να προκαλέσει σημαντικέ βλάβε. Δεύτερον, αποθήκευση των δεδομένων. Στην περασμένη θητεία του Κοινοβουλίου το είχαμε ξανασυζητήσει και είχαμε συζητήσει σε μια συνάντηση διάφορες τεχνολογίες. Και μας είχαν πει ρητά ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος αποθήκευσης. Και βλέπω ότι υπάρχει τελικά. Και εκεί μου δημιουργούνται αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Τα δεδομένα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται. στην αρχή μας είπαν ότι η τεχνολογία αυτή δεν ε, το επιτρέπει, αλλά στην πραγματικότητα αποθηκεύονταν γιατί χρειαζόταν να κάνουν τις επιδείξεις. Άρα πώς τα αποθήκευαν. Τρίτον, πού εντάσσεται το όλο σύστημα στην, ε, στους γενικότερους κανόνες ασφαλείας αεροπλοίας. Οποιεδήποτε, οποιεδήποτε σαρωτές, ακόμα και μεταλλικών αντικειμένων, είναι μία ε, δευτέρ, ε, ε, ελάσσον μέθοδος ε, εντοπισμού τρομοκρατών. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι πληροφορίες για την οργάνωση τρομοκρατικών πράξεων. Αυτές είναι που μας οδηγούν στην, στο, στην εξάρθρωση. γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και προφίλ επιβατών. Τα προφίλ μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Γιατί μια ε, κυρία μεγάλη ηλικία που πηγαίνει ε, διακοπές το καλοκαίρι κάπου σίγουρα δεν αποτελεί κίνδυνο. Μετά, για τα υγρά και τις γέλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνολογία ε, που θα μας επέτρεπε να εξαιρέσουμε αυτά τα ε, προϊόντα από τους ελέγχους και τους κανονισμούς. Θα ήθελα να μου επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει τέτοια τεχνολογία προκειμένου να συμφωνήσω. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, κύριος Μπαχ. Ε, ευχαριστώ για την εργασία που έκανε ο εισηγητής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το θέμα αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ε, ένα κοινό παρανομαστή όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Καταρχήν, ε, η αποθήκευση των στοιχείων. Πιστεύω ότι εδώ αμφισβητείται μόνο το ε, θέμα των εικόνων του σώματος και όχι αποθήκευση δεδομένων, διότι εκεί θα προσκρούσουμε σε προβλήματα προβλήματα, πόσο χρόνο και τι θα αποθηκεύουμε και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ε, όταν μιλάμε για μεσοπρόθεσμη εφαρμογή υπάρχουν πολλές ακτίνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να σκεφτούμε και το προσωπικό. Καταρχήν τους πιλότους και το προσωπικό της ε, καμπίνας ε, που ασχολείται με τους, ε, με τους επιβάτες και να εξετάσουμε και την κοινωνική πτυχή όπως και τη μισθολογική γιατί χωρίς καλό μισθό και καλές κοινωνικές συνθήκες δεν θα υπάρχει προσωπικό το οποίο να είναι άξιο εμπιστοσύνης και να μπορεί να ε, λειτουργήσει και σωστά. Ε, εάν ε, εξετάσουμε και το προσωπικό των τρίτων κρατών θα είχαμε τεράστια προβλήματα και όσον αφορά την πληροφοριακή αλυσίδα όπως απέδειξαν τα παραδείγματα πολλές πληροφορίες έχουν ναι μεν συγκεντρωθεί αλλά μετά δεν μεταδόθηκαν και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Σεναλό για τρία λεπτά. Κυρία Σεναλόβα. Η κυρία Σεναλόβα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και να πω κάτι για την τεχνολογία των ακτινών Χ. Συμφωνώ με αυτούς που ε, είναι κατά της τεχνολογίας αυτής. Θα πρέπει να το γράψουμε αυτό ρητά στην έκθεση. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Μίλησαν για αυτούς τους λόγους συνάδελφοι προηγουμένως. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, διανόμου απαγορεύουν την ε, χρήση ακτίνων Χ για οποιαδήποτε, ε, για οποιοδήποτε λόγο εκτός των ιατρικών εξετάσεων. Οπότε εμείς ε, θα θέλαμε να μην γίνει δυνατή η χρήση ακτίνων Χ. Ορισμένες ομάδες βέβαια έχουν ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο. Θα πρότεινα κάποια εναλλακτική τεχνολογία. Θα προτιμούσα κάποια εναλλακτική τεχνολογία. Αν όμω χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία πρέπει να είναι ασφαλής. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώ ε, να πω, επειδή υπάρχει μια τέτοια ποικιλία. Ε, είχαμε ε, αποφασίσει ε, για τα υγρά την οδηγία και είχε γίνει και μία ακρόαση και κανείς δεν μπόρεσε να μας αποδείξει την αποτελεσματικότητά της και μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσε κανείς να μας πλήσει. Ήταν απλώς ένας καυγάς και ορισμένοι εποφελήθηκαν. Χάρη όμως αυτής της εμπειρίας τώρα μας έχει γίνει μάθημα. Είμαστε σκεπτικιστές, μας, ενδιαφέρονται, ε, ε, μας, ενδιαφέρει το θέμα, αλλά με προσοχή. Κύριε Σέντερ, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντεγκράντες ε, που πραγματικά δείχνει συμβαστικό πνεύμα Συμφωνώ με τον αποκλεισμό της τεχνολογίας των ακτίνων Χ. Πέραν αυτού όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ιδιαίτερως τους ε, ανθρώπους που εκτίθενται τακτικά. Θα πρέπει και να του ενημερώνουμε και να προλαμβάνουμε οποιοδήποτε βλάβη. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, ε, ε, η, και εκεί η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα θα πρέπει να είναι αρμονισμένη η πληροφορία που θα δίδεται. Δεν είναι τον κάθε αεροδρόμιο να το κάνει με το δικό του τρόπο. Αν χρησιμοποιηθούν οι σαρωτές θα πρέπει η ενημέρωση των επιβατών να γίνει με εναρμοσμένο τρόπο. Επίσης ε, χρειάζεται και κώδικα διοντολογία για τους ίδιους εργαζόμενους. Ε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ε, ε αποθήκευσης δεδομένων. Στο, υπάρχουν σκάνερ τα οποία είναι πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία στα οποία όπως αυτό του Αμβούργου καθυστερεί, ε, περιμένεις ε, να ανάψει ένα πρόσημο ε, πράσινο ή κόκκινο φως, κάποιος κοιτάει εκείνη τη στιγμή το, το αποτέλεσμα του σκάν, οπότε είναι σημαντικό να αποφύγουμε τέτοιου είδου προβλήματα. Σε ό,τι διαφορά τα υγρά, σε μια ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ε, είναι σημαντικό να ξαναεκφράσουμε ε, τις αμφιβολίες μας και τις επιφυλάξεις μας παρόλο ότι η προθεσμία του Απριλίου είναι πολύ κοντά. Ευχαριστώ και εγώ ίδιο τώρα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Ντεγκράντες για το έργο σας. Ήσασταν πολύ σχολαστικός. και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να, να ζητήσει κανείς ε, συμβιβασμούς σε ένα τόσο ευρύ φάσμα απόψεων. Συμφωνώ με τον κύριο Μπράτπορτ με την εξαίρεση των υγρών και των γελών. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Έχει δίκιο όμως αυτό που είπε. Πού είναι οι κοινοί κανόνες τελικά. Θα πρέπει να μιλάμε για κοινού κανόνες. στο, όταν πετάει κανεί στο χήθρο, όλα τα παπούτσια θα πρέπει να. Ε, όλοι πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια. Αν όμω πετάξει από το Μάντσεστερ, κανένα δεν σου ζητάει να βγάλει τα παπούτσια σου. Πού είναι η συνέπεια, η λογική συνέπεια μεταξύ αυτών. Ε, ε, αυτό, τα, αυτό το παράδειγμα με τα παπούτσια είναι ένα απλό παράδειγμα, έτσι. είμαι σίγουρος ότι παρόμοια, παρόμοιες καταστάσεις υπάρχουν και σε άλλα αεροδρόμια. Οπότε, ε, το άλλο θέμα, εκτινοβολία εκτείνει χ, είναι προφανέ ότι οι συνάδελφοι δεν συμφωνούν καθόλου. Ε, ούτε και η Επιτροπή ε, Ατομικών ε, Ελευθεριών του Κοινοβουλίου συμφωνεί. Ε, όμως, ε, υπάρχουν κράτη τα οποία δεν βλέπουν να υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της χρήσης των ακτίνων χ. Για παράδειγμα, στη χώρα μου η κυβέρνηση δεν βλέπει πρόβλημα Ο Φίλιπ ε, μας, ε, μας ε, μίλησε για το ίδιο ακριβώ ζήτημα. Χρειάζεται να διδάξουμε και τα ίδια μας τα κράτη-μέλη, να τα πείσουμε ότι είναι σωστή η θέση την οποία συμμεριζόμαστε όλοι εδώ μέσα κατά βάση, σχεδόν όλοι. Πρέπει να πιστούν και τα κράτη-μέλη. Μετά, Λουίσα. Ε, υποστήριξες την ιστορική θέση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα υγρά. Με τις ημερομηνίες του 2011 και του 2013. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει με τα κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή, κρυμμένα πίσω από τη δικαιολογία της ασφάλειας, ε, δεν ε, και κρυμμένα πίσω από ε, το οικονομικό θέμα δεν σκοπεύουν να αγοράσουν μηχανήματα για τον έλεγχο των υγρών. θα πρέπει να μας πει η Κομισιόν τι θα κάνει με αυτά τα κράτη-μέλη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σωστό και θα έπρεπε να φτάσει μέχρι το τέλος Απριλίου. Ε, το transit, οι κανόνες για το transit που έχουμε προβλέψει με την απόδειξη αγοράς βέβαια κλπ. Αλλά όλα να λήξουν το 2013. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Κομισιόν. Η έκθεση είναι περίπλοκη γιατί μπορούμε να κατηγορηθούμε ε, ότι από τη μια μεριά θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και από την άλλη μεριά ότι παραβαίνουμε τις ε, ελευθερίες, ε, τις ατομικές ελευθερίες, οπότε χρειάζεται σολομόντια σοφία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ισορροπία και επιστρέφω στο πρώτο σημείο ο σκοπός είναι να έχουμε κοινούς κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα έπρεπε να επιδιώκουμε. Κομισιόν, κ. Κορνέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συγητή, τον κύριο Ντεγκράντες, για την ε, πολύ σημαντική δουλειά που έκανε στο φάκελο αυτό, στην έκθεση αυτή, ιδιαίτερα τη στιγμή αυτή που η Κομισιόν συντάσσει ε, το δυνητικό μελλοντικό τοπίο στην περιοχή αυτή. Μας βοηθά επίσης ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση στην Επιτροπή επί του θέματος αυτού που θα μας βοηθήσει στο, στην ε, σύνταξη της ε, νομοθεσίας. Υπάρχει αρκετή εμπειρία με τους ερωτές που έχουν εγκατασταθεί εδώ και εκεί στα κράτη-μέλη, το οποίο έχει οδηγήσει και σε αρκετέ τροπολογίε. Ε, θα ήθελα λοιπόν να τομίσω ότι οι σερωτές αυτοί έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά. Σύμφωνα με κανόνες ε, που έχουν αναπτυχθεί τοπικώς. Το έργο που προετοιμάζουμε είναι ακριβώς για να καλύψουμε τα ζητήματα τα οποία έχετε εκφράσει και εσείς, υποβάλει και εσείς, υπό την έννοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως τόνισε και ο κύριος Σίμψον. Γιατί πιστεύουμε και εμείς πράγματι ότι οι σαρωτές είναι μια τεχνολογία πολύ χρήσιμη και πολύ θετική για την ασφάλεια, πολύ καλύτερη από τους ανιχνευτές μετάλλου και θα προτιμούσαμε να μην διατηρηθούν τροπολογίες που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα όπως 67 και τις τεχνολογίες. Αρκετές τροπολογίες αφορούν τις προϋποθέσεις που αφορούν την υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ είναι κρίμα υπό μια έννοια που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ακόμα την ανάλυση αντικτύπου που έχουμε προετοιμάσει, καθότι ακόμα συζητείται εσωτερικά. Όταν θα έχετε τη δυνατότητα να την διαβάσετε, θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που υπευλήθησαν σχετικά με την υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί έχουμε δει ακριβώ τα ίδια θέματα αυτά και πιστεύουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις. Αρκετές λοιπόν τροπολογίε, κατά την άποψή μα δεν θα είναι απαραίτητες υπό το φω των ευρημάτων της ε, ανάλυσης που πρόκειται να έρθει στο φως. Ένα δύσκολο θέμα είναι βεβαίω η τεχνολογία και τα θέματα της εκνοβολίας των ακτίνων. Εδώ ως γενικό κανόνα εκινούμε από το ότι θα έπρεπε να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι υπό την προϋπόθεση ότι η υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται και προασπίζονται. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι, κατα... δεν είναι περισσότερο κατά πόσον πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών φυσικά, αλλά το πώς στην ανάλυση αντικτύπου λοιπόν υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία για την προστασία από ακτινοβολία, οριζόντιας φύσεως και που καλύπτει με ευρύ και γενικό τρόπο το ζήτημα. Γιατί εδώ δεν μιλούμε από μία και μόνο, ένα και μόνο τύπο έκθεσης, αλλά κάθε είδους έκθεση. Κατά πόσον λοιπόν είναι καλύτερο σε αυτήν την νομοθεσία να καλύψουμε το ζήτημα ή στην οριζόντια νομοθεσία έναντι προστασίας προστασία έναντι οποιασδήποτε ευθυνοβολία, δηλαδή. Ε, τώρα για την 168 τροπολογία. Και εμείς βεβαίως θέλουμε να έχουμε επίσημη τοποθέτηση του Συμβουλίου για την προτινόμενη οδηγία, αλλά θα, θα θέλαμε να διακρίνουμε το ζήτημα αυτό, αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ε. απλούστατα γιατί το θέμα της χρηματοδότησης δεν αφορά συγκεκριμένα τους σαρωτές ασφαλείας και αφορά όλα τα μέτρα ασφαλείας. Για τα υγρά, τα αερολήματα και τα τζελ, τις γέλες, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Ντεγκράντης να μην εστιαστούμε τόσο πολύ στην, στην προθεσμία του Απριλίου αλλά περισσότερο να εστιαστούμε στην προθεσμία του 2013 που είναι ο βασικός στόχος που έχουμε και για να απαντήσω και σε ερωτήσει Γκρό ε, και Σίμψον, τι θα κάνει δηλαδή η Κομισιόν. Εφόσον δεν εφαρμόσουν σωστά τα κράτη-μέλη τους κανόνες, αυτή τη στιγμή έχουμε κοινοποιήσει κοινοποιήσεις από αρκετά κράτη-μέλη, τέσσερα προ το παρόν, τα οποία διατίθενται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να ζητήσουμε περισσότερο λεπτομερή εξήγηση του γιατί θα προχωρούν αυτά τα μέτρη για να δούμε και το άρθρο 6 του κανονισμού 300 και κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση εκεί. Και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, θα δούμε κατά πόσον υπάρχει περιθώριο ή λόγος για περαιτέρω διαδικασίες παραβίασης για τα θέματα του φορτίου. Έχουμε αρκετές τροπολογίες εδώ, είναι σημαντικό το θέμα για μας και χαιρόμαστε που καλύπτεται. Το σημαντικό εδώ ζήτημα είναι με το φορτίο το εισερχόμενο και έχουμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες για το εξερχόμενο φορτίο, δηλαδή αυτά που βγαίνουν από την Ευρώπη. Έχουμε Έχουμε 21 και 178 τροπολογίες που αμφισβητούν ίσως κάπως τους ιστορικούς μας κανόνες και αυτές ε, θα θέλαμε να τις δούμε τροποποιημένες για να συμπεριλαμβάνουν και το θέμα του εισερχομένου φορτίου. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Εύα έχει ένα διαδικαστικό. Δεν ήξερα πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, αν θα έχουμε στην απόφαση ή αν θα διατυπωθεί μια νέα πρόταση. Δεν ήταν σαφές. Εγώ υποθέτω ότι θα είναι στην απόφαση. Ε? Δεν θα είναι έτσι. Λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν θέλω να στριμώξω εδώ κανέναν. Αλλά ποια θα είναι η διαδικασία, αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Αν παρακάμψετε, αν η πρόθεσή σας είναι να παρακάμψετε το κοινοβούλιο, το, το, αυτό το green capping θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα red. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σαφές. Αν μιλάτε για τους ερωτές, και όχι το φορτίο, ναι, τους αρωτές λοιπόν, είναι ένα από τα μέσα που είναι στη διάθεσή μας, όπως λέει και ο κανονισμός 300, σύμφωνα και με τη διαδικασία ΠΡΑΚ, έτσι. Είμαστε πάντα εντός του πλαισίου αυτού. Right, Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω για τα δοκιμαστικά αυτά μέσα, καλώς καταλαβαίνω αλλά δεν ξέρω κατά πόσον δίνουμε την εναλλακτική λύση στον ταξιδιώτη, δηλαδή ή θα περάσεις από τις ακτίνες χ ή, θα, ή αλλιώς δεν θα πετάξεις, γιατί αυτό είναι take it or leave it, έτσι. Είναι αναγκαστικό δηλαδή μέτρο, δεν είναι καθόλου εναλλακτικό. Η δοκιμαστική προσπάθεια έχει την ακτή στον αέρα εφόσον τα κράτη-μέλη, οι αρχές τους δηλαδή μας λένε ή θα το κάνεις αυτό ή θα καθίσεις εδώ και δεν θα πετάξεις. Ο κ. Δεγκράντες. Ευχαριστούμε την ε, Κομισιόν που μας διευκρίνησε λίγο τα πράγματα. Να ξεκινήσω με την ε, εξή σχόλιο επί των όσων είπε η Κομισιόν και η κυρία Βιτεμπέργκερ. Ε, εγώ λέω στην γνωμοδότηση αυτή ότι ζητώ νομοθετική πρόταση. Ε, οπότε η δική μου βούληση είναι η συναπόφαση. Αυτή είναι η θέση του εισηγητή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Κομισιόν θα πάρει θέση ούτε πριν ούτε τώρα. Αγώ απλώ ζητώ νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν μέσω αυτή τη νομοδότη πρωτοβουλία. Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώ δεν έκανα λάθο. Δεν έπεσα έξω. Το είχα καταλάβει από τι τροπολογίε και μου το επιβεβαίωσαν οι, ε, οι, οι παρεμβάσει των συνάδελφων. Εντοπίζω σημαντικέ συγκλήσει. Διαφορετική ορολογία, διαφορετική έτσι, προσέγγιση, αλλά τελικά συγκλήσει. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένο. Είμαι αισιόδοξο ε, ότι θα καταλήξουμε σε ε, θετικό αποτέλεσμα. Ο κ. Ε, Φράκριστάιν ε, είπε ότι δεν υπάρχουν να μην ε, υπάρχουν ε, εικόνες, να μην αποθηκεύονται, να μην, χρησιμοποιηθεί, να μην χρησιμοποιηθούν οι ακτίνες ε, Χ και μέτρα για το φορτίο και, το, για την αγροφία μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικά ναι. Ξέρω. Η Air France, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ε, σκύλους στον έλεγχο των φορτίων. Έχω δει τέτοιου είδους ε, μεθόδους και μάλιστα πολύ αποτελεσματικές. Το πρόβλημα είναι με, τη, με τα πρόσωπα, όχι με τα φορτία. Στα φορτία, τα φορτία επιτρέπουν τη χρήση σκύλων. Ε, μετά, για το όνομα. Δεν με νοιάζει. Δεν πρόκειται να το καταστήσω ε, θέμα πρόσκομα. Όχι. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να το προβάλλω ιδιαίτερα. Κυρία Μέισνερ, να, ε, κα, να απαγορευτούν οι εκτενές Όχι, αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή μέθοδος. Μπορούμε να ζητήσουμε να απορριφθεί ως μέθοδος, αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω τη λέξη απαγόρευση. Στην ε, πραγματικότητα όμως συμφωνούμε, έτσι. Τροπολογία 29. Λέτε ότι είναι καλή. Να χρησιμοποιηθούν και, σε, να χρησιμοποιηθούν και, άλλες, και άλλοι τρόποι ανείχνευσης. Ωραία. Συμφωνώ, εγώ σας είπα. Είδα τα σκυλιά στη Γαλλία και μου φαίνεται πολύ αποτελεσματικό σύστημα. Πολύ ε, τάχιστα αναλύονται, ε, αναλύεται μεγάλος αριθμός ε, εμπορευματοκιβωτίων και containers και τα σκυλιά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και στις επιδείξεις και στην πράξη. Μετά, ε, για τις ακτίνες χ έχω να πω και το εξής. Ο εισηγητής πρέπει να ενημερώνεται. Ε, υπάρχουν ορισμένες ακτινοβολίες χ οι οποίες σύμφωνα με τους τεχνικούς, με τους εμπειρογνώμονες, είναι διαφορετικές, διαφορετική από ότι άλλες που πραγματικά εκπέμπουν βλαβερές ακτινοβολίες, που είναι βλαβερές ακτινοβολίες. Εγώ παρόλα αυτά δεν κάνω διάκριση. Δεν κάνω διάκριση ανάμεσα σε διαφορών ειδών ακτίνες χ. Γι' αυτό το λόγο λέω να μην χρησιμοποιούνται. Συνεπώς δεν κάνω διακρίσεις, ας μην συζητήσουμε για αυτό το θέμα, έτσι. Προστασία δεδομένων. Συμφωνούμε. Οπότε πολύ σωστά όσα είπατε, δεν έχουν να πω τίποτα. Κύριε Φώστερ. Και ο κύριος Μπράντμπορ και η κυρία Φώστερ. Ε, ο κύριος Μπράντφορντ έφυγε, λυπάμαι. Ε, είναι ομός ο κύριος Μπράντφορντ πολύ συχνά. Ε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι λογική η στάση τους. Γιατί από τη μια μεριά υποστηρίζουν την ε, επικορικότητα και από την άλλη μεριά λένε να υποχρεώσουμε όλους, να υποχρεώσουμε όλους. Ε, δεν γίνονται αυτά τα δύο μαζί. Γιατί σε τέτοιου είδους θέματα ξεκινούν οι νομές Πολιτείες και μετά τα ξαδελφάκια τους και δεν ρωτάνε κανέναν. Και τα υγρά μας τα επέβαλαν και τα μέτρα αυτά μας τα επιβάλλουν. Οπότε θα πρέπει και τα κράτη και οι επιβάτες να έχουν ελευθερίες. Απ' την άλλη μεριά συμφωνώ, κοινοί κανόνε. ναι. Αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Όποιο εφαρμόζει τα μέτρα που θέλει, όποια είναι και αυτά στο πλαίσιο τη ελαστικότητα, θα πρέπει να τηρεί παρόλα αυτά του κοινού κανόνε, Το ελάχιστο. Μετά, η κυρία Φώστερ λέει, ε, συμφωνεί με τα... Ε, ε, να, να μην χρησιμοποιούμε ε, προφίλ. Απ' την άλλη μεριά, άλλοι συνάδελφοι θέλουν προφίλ. προφίλ. <laughs> Ρητά. Οπότε είναι δύσκολο να ε, τα συμβιβάσουμε αυτά. Και ταυτόχρονα η κυρία Φώστερ μίλησε για αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία ακτινών χ που χρησιμοποιείται στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, και που λένε ότι είναι βραβερή. Τέλο Κυρία Βίλς, υπέρ το, της έκφρασης ε, να προστατεύουμε την υγεία και βέβαια να διασφαλίζουμε τα δεδομένα πολύ σωστά. Ποιος Γκρός μας υπενθύμισε την επικορικότητα, την πραγματική σου επικορικότητα. Αυτή τη στιγμή γίνονται ε, πειραματισμοί σε διάφορα κράτη-μέλη και με, ε, εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους. Ανεξάρτητα από το τι θα πούμε εμείς όμως, τα κράτη-μέλη πάντοτε θα έχουν την νομική δυνατότητα να εφαρμόσουν συστήματα πιο αυστηρά. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το απαγορεύσουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Μπαχ, συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Συμφωνώ και με τους επόμενους ομιλητές. Κυρία Γιάλα, μίλησε για τα ευάλωτα άτομα. Το θέμα το έχω ήδη συμπεριλάβει στην έκθεση. Όμως βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν να ξεκαθαριστεί ακόμα περισσότερο. Να, μην, να γίνει σαφές ότι δεν μιλούμε μόνο για τα παιδιά, τους ασθενείς κλπ. αλλά και τους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται πολύ συχνότερα ε, σε τέτοιου είδου συστήματα. Μετά, κύριε Σίμψον, είπατε κι εσεί, μιλήσατε για του κανού κανόνε. Και εγώ το ίδιο λέω. Μιλώ για ελάχιστε προδιαγραφέ. Και εσεί είπατε όχι στι ακτίνε Χ, καμία διαφωνά. Να, άλλη μεριά, είπατε ότι θέλουμε, θέλει ε, να διατηρήσουμε τις ημερομηνίες της 29 Απριλίου και του 2013. Κομισιόν συμφώνησε με αυτό που είπα, παρόλο που δεν ήμασταν συνεννοημένοι. Αφόσον εμεί θα πάρουμε αποφάσει, δηλαδή θα εκδώσουμε αυτή την γνωμοδότηση μετά τι 29 Απριλίου, γιατί να μιλήσουμε για τι 29 Απριλίου. Α ε, ενώσουμε τι δυνάμει μα για το 2013. Γιατί να μιλάμε για πράγματα τα οποία ήδη θα έχουν αποφασιστεί όταν εκδοθεί η γνωμοδότησή μα. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την υποστήριξή της και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση επιπτώσεων, γιατί αυτή η αξιολόγηση θα μας δώσει αποτέλεσμα για το πώς πήγαν τα, οι και θα μπορέσει να μας διαφωτίσει για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, σύγκληση και συνένεση και είμαι σίγουρος ότι ε, θα υπερψηφιστεί αυτή η γνωμοδότηση, όχι επειδή την έφτιαξα εγώ, αλλά επειδή συμφωνούμε κατά βάση. Ευχαριστώ κύριε Τιγκράντης. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα είναι το Μάιο και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Με, ε, συγχωρείτε. Επιτροπή λοιπόν Μάιος και Ορμέλεια Ιούνιος. Επόμενο σημείο. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ε, συνδυναμικός χώρος παρουσίαση ε, από τα δύο σημειώματα που είχαν ζητήσει και οι συντονιστές ε, μεταφορικών που είχαν ζητήσει μετά την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας της εισηγήτριας κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ιανουαρίου και επί τη βάση εγγράφων υφισταμένων θα παρουσιάσουν την κατάσταση και τον αντίκτυπο για την, για την διάκριση των ε, ρυθμιστικών ε, φορέων σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τους πόρους στα συνδρομικά σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η Steer Davis Gleave έχει ολοκληρώσει το έργο αυτό και θα το παρουσιάσει τώρα από έναν από τους βασικούς ε, συνεργάτες, τον κύριο Φρανσίσκο Διανόρη, οπότε σας δίνω αμέσως το λόγο για να πάμε μετά στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλλον θα έχετε λάβει αντίγραφα της παρουσίασης ε, έντυπα, γιατί μάλλον θα είναι πιο εύκολο έτσι από ότι με προβολή στην οθόνη. Λοιπόν, όπως είπε ο Πρόεδρος, ε, μας είχε ζητηθεί να δούμε δύο διαφορετικές μελέτες. Μία για το unbundling, unbundling και μία για, τις, ε, για τα ρυθμιστικά σώματα. Και θα σας κάνω μία σύντομη εισαγωγή για το τι είναι οι δύο αυτές ε, μελέτες. Μία επισκόπηση της, γενική επισκόπηση της αγοράς για τα δύο σημειώματα αυτά και μετά μία σύντομη συζήτηση για τα ίδια τα σημειώματα. Έχουμε την υπολογία λοιπόν και δομή των ρυθμιστικών φορέων και αντίκτυπος της διάκρισης μεταξύ της διαχείρισης του ε, εξοπλισμού και των μεταφορών. Έχουμε διαφορετικά πρότυπα και μοντέλα για τη διάκριση αυτή στα διάφορα κράτη-μέλη, σύντομη σημείωση. Εδώ έχουμε σημειώματα και όχι λεπτομερείς μελέτες. Ω εκ τούτου δεν έχουμε δει τα πάντα σε κάθε λεπτομέρεια σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτώντα τώρα σύντομα την αγορά και που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα συνδρομικά. Καταρχά, μεταφορά επιβατών από το 2000. Η συμμετοχή είναι περίπου στο 60% για του σιδηροδρόμους τα τελευταία χρόνια. Θα δείτε και ένα γράφημα το οποίο όμω ε, δεν δείχνει τις αμαξοστοιχίες, δεν συμπεριλαμβάνει τις αμαξοστοιχίες, είμαστε περίπου στο 73%. Έχει υπάρξει σημαντική αύξηση σε κάποια κρατημέλη, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, αλλά στις, ε, στα ασπάνω αντίγραφα είναι το, το τρίτο από την αρχή Υπάρχουν, έχουν υπάρξει κάποιε διακυμάνσει, αλλά δεν έχει αλλάξει η συμμετοχή σε σημαντικό ποσοστό. Η συμμετοχή λοιπόν στην αγορά, η παρουσία στην αγορά, είναι κάπως ευρύτερη, αλλά όχι σημαντικά ευρύτερη στην αγορά των επιβατών. Κάπου πάνω από το 10%. Σημαντική αύξηση σε κάποιες αγορές όπω Λετωνία, Αυστρία και Γερμανία, αλλά συνολικά το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σταθεροποιηθεί σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς. Μιλώντας για την συμμετοχή στην αγορά, βλέπουμε μια διαφάνεια με την εξέλιξη της αγοράς εμπορευμάτων, της μεταφοράς εμπορευμάτων. Μπορείτε να δείτε ότι έχουμε κάποιες πολύ, κάποια πολύ ψηλά μεγέθη στο Ηνωμένο Βασιλείο, την Εστονία, τη Δανία και την Πολωνία, αυτό που δείχνει αυτό είναι ότι κατά μέσον όρο είχαμε μια αύξηση των συνδραμικών επιχειρήσεων μέχρι το 22% στο 2009 είχε φτάσει αυτό. Με κάποιες υψηλές καμπές αύξηση στην Εστονία για παράδειγμα και στην Αυστρία Τα έτη που έχουν επιλεχθεί έχουν βασιστεί σε προηγούμενες μελέτες, όπως είχε πει και ο Πρόεδρος 2005 και 2006 σε άλλες μελέτες του Steve Glavis, Davis Gleave και τα τελευταία στοιχεία προκύπτουν από την ίδια την έκθεση της Κομισιόν RMMS. Πάμε τώρα στις ρυθμιστικές αρχές. Μια μικρή εισαγωγή. Ο βασικός στόχος είναι να εξασφαλίζουν μια ισότιμη ε, διαχείριση της αγοράς σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή να αποκλείονται οι διακρίσεις. Το άρθρο 30 της οδηγίας απαιτεί να είναι ανεξάρτητες οι αρχές αυτές από την ε, διοίκηση των συνδρομικών επιχειρήσεων όπως και από τις αρχές κατανομής πόρων. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στην αδιατύπωση για την εντολή και την ισχύ των αριθμιστικών αρχών ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος τους, να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες εξάρτητα και εξπόστ. Για παράδειγμα σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο της διαχείρισης υποδομών, όπως και για να τις έχουμε ως επιμέρους αρμόδια αρχή σε, σχέση, σε σύγκριση μάλλον προς τις υπόλοιπες αρχές που μπορεί να υπάγονται στο αρμόδιο Υπουργείο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Τα είδη τώρα των εθνικών αρχών διαιρούνται σε δύο τομείς. Το πάνω μέρος που βλέπετε στην σελίδα έχουμε τις επιμέρους και τις ενσωματωμένες αρχές. Τι σημαίνει αυτό το stand alone δηλαδή επιμέρους. Πρόκειται για καθαρά στη δυναμική αρχή, ενσωματωμένη είτε ευρύτερα σε μεταφορικό φορέα, φορέα μεταφορών, ή ακόμα ευρύτερο σε σχέση με, για παράδειγμα, αρχές ανταγωνισμού. Οι περισσότερε αυτή τη στιγμή είναι επιμέρους αρχές. Υπάρχουν και υπέρ και κατά. Και στη μία και στην άλλη κατεύθυνση για τις δημιουργικέ αρχές σχετικά με την εστίαση που κάνουν είτε μόνο στους ιδεοδρόμους είτε αν έχουν μια ευρύτερη εικόνα της αγοράς ε, και τα λοιπά. Υπάρχουν πλέον εκτίματα σε μια προσέγγιση ενσωμάτωσης, όπου υπάρχει ένα ενιαίο ε, γραφείο ε, ανάλυσης κόστους, για παράδειγμα, αλλά και οι δύο αυτές προσεγγίσεις συμμορφούνται προς τις προϋποθέσεις οδηγίας. Στο κάτω μέρος της προβολής αυτής βλέπουμε τι προϋποθέτει η αναδιατύπωση ιδιαίτερα του το άρθρο 5 με διαίρεση μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι απολύτως ανεξάρτητες από Υπουργεία και αυτές που είναι συνδεδεμένες κατά κάποιο τρόπο σε Υπουργική Αρχή. Εδώ η διαίρεση είναι πάνω κάτω η ίδια. Και αυτό συζητούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια και στο σημείωμα. Τώρα βλέποντα τη δομή και τα, τους τύπους των εθνιστικών αρχών και κά, κατά κάποιον τρόπο την αποτελεσματικότητα είδαμε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές. Η πρώτη από τις οποίες είναι οι παραβάσεις που έχουν ε, ε, καθοριστεί από την Κομισιόν και όπως φαίνεται υπάρχουν αρκετές τέτοιες σε σχέση με αρκετά κράτη-μέλη. Ανεπαρκής ανεξαρτησία από τις ιδεονομικές επιχειρήσεις ε, και τη διαχείριση των υποδομών ή από τις αρχές ανταγωνισμού σε αρμοδιότητες ε, επιβολής του, του νόμου και των κανονισμών. Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο για λεπτομερή απόφαση. Ιδιαίτερα Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία και Ισπανία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνιστικές ακριβώς αρχές ε, και αυτή εδώ η διαφάνεια, ο πίνακα αυτό κοιτάει απλώς τις παραβάσεις σε σχέση με ρυθμιστικές αρχές και όχι τις συνολικές παραβάσεις. Επίσης έχουμε συγκρίνει τη συμμετοχή των νεοεισερθόντων εταιριών επιχειρήσεων σε σχέση με τις περιπτώσεις παραβάσεων ή μη παραβάσεων. Υπάρχουν όμως χώρες με υψηλότερες συμμετοχές αγορές που έχουν χαμηλότερο επίπεδο παραβάσεων. Που είναι μία από τις συγκριτικές μελέτες που είχαμε και στο σημείωμα. Κάτι που συχνά τίθεται από τους ενδιαφερομένους ε, τον κλάδο συνολικά Στι που είχαμε μαζί τους είναι η διοικητική ικανότητα κάποιων από τις ρυθμιστικές αρχές αυτές, όχι σε όλο το φάσμα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις έχει διατυπωθεί συγκεκριμένη ανησυχία. Εμείς σημειώνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις αρχές έχουν προσωπικό κάτω των 60 ατόμων. Και δυνητικά, ο αριθμός αυτός των υπαλλήλων αδυνατεί να διαχειριστεί το σύνολο της αγοράς, όπως σημαίνει με την Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή. Με αγορά 25 επιχειρήσεων ε, ε, εμπορικών μεταφορών και άνω των 50 υπολείπων επιχειρήσεων μεταφορών. Αδυνατούν λοιπόν να δουν το, το σύνολο του φάσματος των προβλημάτων και των, των προβληματικών σημείων που μπορούν να ανακύψουν σε όλη αυτή την αγορά. Άλλη μια ανάλυση που, στην οποία προχωρήσαμε ήταν μια απλή δοκιμή για να εξετάσουμε κατά πόσον υπήρχε πραγματική ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αυτών αρχών. Οι πρώτες τρεις στήλε είναι αυτή η απλή δοκιμή που σας λέω, δηλαδή κατά πόσον το Υπουργείο έχει την, το απαραίτητο γραφείο με την, στο, στο ίδιο σημείο με την ρυθμιστική αρχή, τι γίνεται με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, αν υπάρχουν ε, επικαλύψεις με, την, ε, με τον οργανισμό διαχείρισης της υποδομής και τον οργανισμό διαχείρισης των μεταφορών, όπως και για τη χρηματοδότηση. Γιατί από μόνο του αυτό είναι ένα στοιχείο ε, που μας δείχνει το επίπεδο ανεξαρτησίας, αν θέλετε. Αλλά σχετικά με αυτό υπάρχουν, έχουν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες. Συνοψίζοντας λοιπόν, πού οδηγούμε θα έχουμε δει την αποτελεσματικότητα σε ένα φάσμα πανευρωπαϊκό για το οργανωτικό του μοντέλο, την χρηματοδότηση, του πόρου, το προσωπικό. Σίγουρα πρέπει να ισχυθεί η φυστάμενη νομοθεσία για να εξασφαλίζει την ε, ανεξαρτησία την πιο αυξημένη των ρυθμιστικών αρχών και θα πρέπει να έχουν ε, του απαραίτητου πόρου και να μπορούν να δρουν γρήγορα, ταχαίω, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Οι ρυθμιστικέ αρχέ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε από τι κυβερνήσει, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άμεσο συμφέρον κυβερνητικό για μια επιχείρηση σιδηροδρομική ή διαχείριση υποδομή. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι και η απαραίτητη αρμοδιότητα να έχει το συνολικό έλεγχο επί των επιχειρήσεων η ρυθμιστική αρχή και αυτό ποικίλει από κράτο σε κράτο μέλο. Προχωρώντας τώρα στο σημείωμα για την ε, διάκριση, στην οποία είχα αναφερθεί, προφαλώς έχουν, ε, έχουμε προχωρήσει και σε, άλλες, σε άλλα είδη διάκρισης, σε άλλους τομείς δηλαδή, πάντα ακούμε ότι η σιδηρόδρομη είναι διαφορετική Σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί και να αληθεύει αλλά παραμένουν ουσιαστικότατα προβλήματα για τεχνολογικά εμπόδια, διαλειτουργικότητα κτλ. Η Κομισιόν έχει ήδη πει σαφέστατα και το Κοινοβούλιο το έχει επιβεβαιώσει αυτό μέσα των οδηγιών ότι θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητα ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε επιχείρηση τηλεδρομική για την κατανομή των πόρων. Υπάρχουν πλεονεκτήματα λοιπόν και μειονεκτήματα της διάκρισης αυτής, του διαχωρισμού αυτού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σημείωμα και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον κατακόρυφο αυτό διαχωρισμό με διαφορετικό αντίκτυπο επί του ανταγωνισμού κάθε φορά. Τα διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν ε, επιλέξει διαφορετικές προσεγγίσεις ε, επί τη βάση των μελετών από την Κομισιόν. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες ως, σε σχέση προς το διαχωρισμό όπου η αρχή διαχείρισης του υποδομής είναι διαφορετική από την αρχή διαχείρισης των μεταφορών ή όταν έχουμε νομικά διάκριση αλλά στην πράξη έχουμε ανάληψη δραστηριοτήτων που ε, επικαλύπτουν τις δύο διαχείρισεις της υποδομής δηλαδή και τις μεταφορές ή έχουμε θηγατρικές επιχειρήσεις που πάλι καταλήγουν στην ίδια επιχείρηση και έχουμε μια ε, de facto ενσωμάτωση αν θέλετε, συγκέντρωση και όχι διαχείριση. Και πάλι εξετάσαμε διάφορους τομείς. Καταρχήν η μελέτη της Επιτροπής ε, εξέτασε τις διάφορες κατηγορίες που προανέφερα και ουσιαστικά ε, εξέτασε τα κράτη-μέλη ε, την κατάσταση που αντικατοπτρίζεται το 2009. Βεβαίως είναι μια ρευστή κατάσταση η οποία αλλάζει συνεχώς και ενημερώνουμε την πληροφόρηση ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, καταλήξει ότι ε, το, τα τρέχοντα πρότυπα δεν συνάδουν με την εφαρμογή του πακέτου. Και όσον αφορά την ανάλυση που είχε ξεκινήσει ο Steve David ε, Cleave εξετάζοντας τον βαθμό ανεξαρτησίας και ορισμένες ε, δοκιμές τις οποίες είχαμε κάνει εκείνη την εποχή ε, κατέληξαν ε, ότι τα στοιχεία έπρεπε να ενημερωθούν σε επίπεδο των κρατών μελών και βλέπετε εδώ ένα συνοπτικό πίνακα που παρουσιάζει αυτά τα οποία έλεγε η έκθεσή μας σχετικά με τη διάταξη. Αν δηλαδή όλοι ε, οι στο ίδιο κτίριο γραφείων, αν ε, υπήρχε καταμερισμό ρυθμός των περιουσιακών στοιχείων λοιπά. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τον πίνακα αφό, αλλά όσο περισσότερα ναι υπάρχουν, τόσο περισσότερο ανησυχούσαμε εις ε, το, ε, στην ανάλυση αυτή. Γι' αυτό και διατηρήσαμε τα στοιχεία αυτά στο σημείωμά μας, διότι είδαμε ότι υπήρχαν και άλλοι τομείς ότι ορισμένοι δηλαδή ε, διευθυντές υποδομών προστάτευσαν ε, τα γραφεία που τους είχαν ανατεθεί και υπήρχαν και άλλες δοκιμασίες που μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τα θεσμικά όργανα, με τα έγγραφα αλλά στα μέτρα που θεωρούμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη σημαντικά. Όλοι γνωρίζετε πόσο προχώρησαν οι παραβιάσεις και δεν θα σταματήσω σε, αυτό το, σε αυτή τη διαφάνεια αλλά βλέπετε ότι δεν υπήρχε επαρκής εξασφάλιση των ε, διευθύνσεων υποδομών και της σωστής κατανομής. Στο σημείο με αυτό δείχνουμε και πέντε μελέτες περιπτώσεων που ήταν μία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και αναφερόμαστε στα πρότυπα τα οποία συζητήσαμε προηγουμένα, δηλαδή μία τελείως ολοκληρωμένη μονάδα και είδαμε ότι στην ε, μειοδότηση ε, υπήρξαν ε, αυξήσεις σημαντικές των εξόδων μετά το 2000 για διάφορους λόγους και ορισμένες από αυτές τις αυξήσεις δαπανών ήταν υπερβολικές σε σχέση με τη συρρήκνωση του επιχειρησιακού πλαισίου και ιδίως σε σχέση με τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχαμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, είχαν αποκλειστεί ε, επενδύσεις οι οποίες ήταν μειωνόμενες δαπάνες και στην ε, Ολλανδία διατυπώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία σαφής απόδειξη ότι αυξήθηκαν οι οι δαπάνες και ο διαχωρισμός βελτίωσε την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Στην Ιταλία είδαμε ότι ε, υπήρξε διείσδυση στην αγορά εμπορευμάτων και οι ε, νέοι ε, εμπλεκόμενοι συνέχισαν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους χωρίς να υπάρχει μία απόδειξη αυξήσεως Στη Γαλλία ε, είδαμε ότι ε, ε, καθυστερεί ο ανταγωνισμός και περιορίζεται η δυνατότητα εισόδου της GDI. Όσον αφορά την αποκέντρωση Ε, ε, συμπεριλάβαμε και τον δίκτυ ε, αποδεσμεύσεως και σε ποιο τομέα ή σε, ποιο βαθμό είχαν προχωρήσει στο 2007 σε σχέση με άνοιγμα της αγοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη την ε, τον διαχωρισμό και ε, το ποσοστό της αγοράς των μη εμπλεκομένων βλέπουμε ότι υπάρχουν αγορές με πολύ μεγάλο ποσοστό της αγοράς σε μη εμπλεκόμενους και συγχρόνως ε, υπάρχουν και ολοκληρωμένα πρότυπα οπότε δεν μπορούσε κανείς να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα βάσει αυτών των στοιχείων και κατά λίγο τώρα στα συμπεράσματά μου ότι υπήρξαν δομικές αλλαγές και ουσιαστικά οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων παραμένουν και ε, θα υπάρξει μεγαλύτερος διαχωρισμός της διαχειρήσεως της υποδομής και ε, των χρηστών και θα πρέπει ε, ε, να εξετάσει κανείς εάν μπορούν να συγκατοικήσουν οι διάφοροι παράγοντες κατά τρόπον ώστε να εξεταστούν οι διάφορες εναλλαστικές ε, λύσεις ε, και να λειτουργήσουν ουσιαστικά, αν όχι νομικά, ε, αν θα χρειαστούν δηλαδή συντονισμοί του προγράμματος, ε, πληρωμή ποινών για καθυστέρηση και ούτω καθεξής διαπιστώσαμε επίσης τάσεις στα έξοδα και τις τιμές και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον ομιλητή για την παρουσία της εκθέσεώς του, αλλά θα ήθελα τώρα να σας πω ότι δεν συζητάμε την έκθεση Σαρικιάνη ουσιαστικά, ούτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι αυτό ε, θα γίνει με την υποβολή των τροπολογιών στις 20 Ιουνίου ε, εξετάζουμε αυτήν την έκθεση. Όσοι λοιπόν ξεκινάει να, ε, αλλάζει θέμα θα επαναφέρεται άμεσα στην τάξη. Και πρέπει να σας πω ότι έχω 150 ομιλητές Οπότε ο καθένας θα πρέπει να μιλήσει δύο λεπτά. Διότι διαφορετικά, εάν δεν σας ικανοποιεί, πρέπει να σας πω όπως έχω επαναλάβει, ότι δεν ελέγχω το χρόνο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον, στον ομιλητή, δηλαδή στην κυρία Σαρεκιάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πραγματικά για την ε, παρουσίαση των briefing notes, όπως είπε και ο Πρόεδρος Προφανώς δεν πρόκειται για μελέτες ε, που πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχέστερα, αλλά για την ε, παρουσίαση, την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης. Πάντως και σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές αρχές και την πρόταση διαχωρισμού διάκρισης, είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που προκύπτει από διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση με τις ε, οδηγίες της πρώτης δέσμης της σιδηροδρομικής. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει καταρχάς ε, μετά από αυτήν την εισαγωγή είναι δύο διευκρινήσεις που θέλω να υποβάλω στον ε, κύριο Διονόρη αφαιρώ, αφενός το σύστημα του διαχωρισμού. Θα ήθελα να καταλάβω αν κατά την άποψή σας έτσι όπως εσείς το μελετήσατε το θέμα τα συστήματα αυτά δηλαδή όπου έχουμε την, ε, δηλαδή συστήματα που έχουμε τη διάκριση και άλλα συστήματα που έχουμε μερική ή καθόλου διάκριση Υπάρχουν δύο σημεία λοιπόν που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον μου. Το γερμανικό σύστημα θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικό, γιατί αυτό θα μας επέτρεπε να κάνουμε κάποιες ε, αξιολογήσεις σε σχέση με ε, άνοιγμα της αγοράς, με κίνηση τον διαχωρισμό ή όχι. Και το άλλο είναι το Ολλανδικό σύστημα, σε σχέση με κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας, ε, κοστολόγησης και σύστημα το οποίο λειτουργεί και με μειωμένο κοινωνικό κόστος και με την ανταπόκριση που δίνει, την, κάλυψη που δίνει στον επιβάτη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονες που μας διέθεσαν τα στοιχεία διότι η Λευκή Βίβλος ε, ήταν ε, σαφής ως προς την, τον διαχωρισμό των υποδομών και ε, γι' αυτό βλέπουμε ότι ε, στηρίζεται η άποψη αυτή ιδίω όσον αφορά το unbundling ε, είναι κάτι το οποίο να αποδεικνύουν και οι εμπειρογνώμονες αλλά αν δούμε κατά πόσον διαχωρίζεται η, διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις εάν αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό εάν αυξάνει το Βλέπουμε ότι στην Ιταλία δεν προχώρησε το θέμα. Για τη Γαλλία δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Καλό θα ήταν να έχει εξεταστεί και η γερμανική περίπτωση σύμφωνα με τον δίκτυ IBM διότι βλέπουμε ότι καμία ανάλυση εδώ δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την Ανατολική Ευρώπη και για το πώς προτίθενται ε, ε, να ανοίξει η αγορά σε αυτές τις χώρες. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε μία πλήρη, ένα ε, πλήρες unbundling σε διάφορες χώρες, τότε το, το, κράτης, το κράτος παραμένει 100% μέτοχος και στη χρηματοδότηση και το προσωπικό, τι μας ενδιαφέρει πώς επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Έπρεπε να δούμε τι γίνεται. Ε, όσον αφορά τα regulatory bodies, όντως ε, αυτά πρέπει να είναι τελείως ε, ανεξάρτητα από τη διαχείριση των υποδομών και από την διεκπαιρέωση των καθηκόντων και όπως γίνεται στη Γερμανία παραδείγματος χάρη είναι σωστό να υπάρχει διαχωρισμός των διαφόρων λειτουργών λειτουργιών και γενικώ θα συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό. Εδώ υπάρχει μία πρώτη πρόταση, αλλά με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν είχα δει το όνομά σας. Κύριο Στρεμόσα. Καταρχήν, έχω προβλήματα με τη διαδικασία αυτή τη αναδιατύπωση. Την περασμένη εβδομάδα πήραμε αυτά τα δύο ντοσιέ, τα briefing notes, μόνο στα αγγλικά. Πολλοί από του ε, συναδέλφου δεν τα έχουν καταφέρει να τα, να τα διαβάσουν. Συνεπώ, θα ήθελα να ζητήσω από την Γραμματεία επαρκή χρονική, ε, χρονική περίοδο για την υποβολή τροπολογιών και για τη μετάφρασή του. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική αρχή, το ρυθμιστικό φορέα, όταν διάβασα αυτό το έγγραφο, ε, επιβεβαιώθηκε αυτό που είχα υπόψη μου, ότι ε, ένας ισχυρός ε, ρυθμιστικός φορέας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το άνοιγμα των αγορών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Οι χώρες που έχουν πιο ανοιχτές αγορές είναι αυτές που έχουν ε, του πιο ισχυρούς ε, ρυθμιστικούς φορείς ε, με το επαρκές προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση. Η Γερμανία και η Ηνωμένο Βασίλειο από τη μία μεριά και η Ισπανία, η Ιταλία από την άλλη. Είναι ο, η βασική βασικό όρο ε, έτσι ώστε η πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο να γίνεται χωρί διακρίσει. Συνεπώ, οποιαδήποτε νομοθετική πράξη θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ρυθμιστικοί φορεί θα έχουν επαρκέ προσωπικό και επαρκή, αρμοδιότητε και χρηματοδότηση. Επίση, οι αποφάσει των ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα, και μάλιστα θα μπορούσε να λαμβάνεται ε, πιο ε, γρήγορα η απόφαση αν είχαμε και ένα ευρωπαϊκό επίπεδο ρύθμισης. Ευρωπαϊκό επίπεδο ρύθμισης μόνο για τις ε, περιπτώσεις που οι εθνικοί φορείς, ε, οι εθνικοί φορείς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έχοντας διαβάσει το έγγραφο για τον διαχωρισμό ανάμεσα στο μεταφορικό έργο και τη διαχείριση των υποδομών, ε, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο διαρθρωτικό μοντέλο και το άνοιγμα των αγορών. Έχουμε χώρες που έχουν ανοιχτή αγορά με χωριστά μοντέλα, όπω οι κάτω χώρε και το Ηνωμένο Βασίλειο, και έχουμε και ανοιχτέ ε, αγορές με εν μέρη διαχωρισμένα συστήματα όπως η Αυστρία και η Γερμανία. Και δεν υπάρχει επίσης σχέτιση ανάμεσα στο ε, μερίδιο αγοράς που έχουν οι, οι, οι παραδοσιακές ε, και στο ε, σύστημα, στο μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στο μοντέλο αποσύνδεσης. Συνεπώς, θα χρειαζόμαστε ανεξάρτητα ισχυρά, ανεξάρτητους ε, ισχυρούς ρυθμιστικούς ε, φορείς με επαρκές προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση για να ε, δίνουν απάντηση σε οποιασδήποτε ε, προσφυγές γίνονται. Και χρειαζόμαστε για την περίπτωση που αυτά δεν λειτουργούν ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Είναι ατυχές ότι έχουμε δύο λεφτά μόνο μετά από όλη αυτή τη μακριά παρουσίαση που δεν είδα κανένα νέο στοιχείο και κατακρίνω ότι δεν περιελήφθησαν περισσότερα κράτη, ότι απεκλείστη η Γερμανία που είναι το μεγαλύτερο κράτος και επιπλέον ε, θα μας αν η διαφορά των αριθμών μεταξύ της ε, Γερμανίας και της Γαλλίας διότι έχουμε μία ε, εξέλιξη μείον 55% στη Γαλλία και συγχρόνως μια μεγάλη αύξηση στη Γερμανία. Αυτό άξιζε να ερευνηθεί. Στην ε, Εσθονία παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι προχωρούν οι ιδιωτικοί σιδηρόδρομοι ενώ στη Σλοβακία υπάρχει μία μείωση και φαντάζομαι ότι εκεί το, το, το κόστος ε, των διοδίων είναι τόσο ψηλό ώστε γι' αυτό δεν υπάρχουν οδικές μεταφορές. Αυτό θα έπρεπε να έχει εξεταθεί και να δούμε ποιοι είναι οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο. Διότι κατ' εμέ αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι το unbundling αλλά τρεις διαφορά. Το regulatory body που πρέπει να είναι καλά επανδρομένο γιατί αν στην Ιταλία έχουμε 10 ανθρώπους και πρέπει να κάνουν τη δουλειά που σε άλλα κράτη κάνουν 100 άτομα δεν μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα και ε, μέχρι να έχει κανείς ένα σλότ ε, θα έχει καταρρεύσει η σιδηροδρομική εταιρεία γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Επίσης ε, στη μία χώρα μπορεί να παίρνει κανείς στη Γερμανία αποφάσει σε λίγες μέρες και στη Γαλλία περιμένει δύο χρόνια και να μην λαμβάνει καμία απάντηση. Τέλος πώς κατανείμονται οι πόροι. Και τρίτον όπως είπα το unbundling δεν μας ενδιαφέρει, είναι και άλλα που μας ενδιαφέρουν όπως το regulatory body και θα ήθελα να έχω την απάντηση από τους γαλλικούς και τους γερμανικούς συνδυροδρόμους γιατί περισσότερα ερωτήματα μου δημιουργήσατε. Ήθελα να ρωτήσω τον παρουσιαστή μας δύο ερωτήσεις. κοιτάζω αυτή την αναμόρφωση ε, με ένα στόχο μόνο, να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και να μειώσουμε το κόστος της μεταφοράς ε, εμπορευμάτων και εδώ διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει επιτευχθεί. Δηλαδή οι περισσότεροι από εμά θα ήθελαν να δουν ε, όχι μόνο να ανοίξει η αγορά αλλά να εμπλακούν και ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εσείς βλέπετε ένα τέτοιο συσχετισμό. Ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο διότι δεν μας είπατε ε, τι γίνεται. Οι τρεις χώρες της Βαλτικής και η Φιλανδία έχουν ένα ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό σύστημα και το σύστημα των σιδηροτροχιών τους είναι πιο φαρδί. Πιστεύετε λοιπόν ότι για να υπάρξει διαχωρισμός οι εταιρείε Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έχουν καλή μεγαλύτερες δυνατότητες και θα υπερτερήσουν των σοβιετικών εταιριών. Ε, εσείς σαν εισηγητής μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε 5-10 λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στους επόμενους ερωτώντους. Αλλά ουσιαστικά γιατί η Γερμανία απεκλείστη από το, τη μελέτη και γενικώ έχετε το λόγο για 5-10 λεπτά να δείτε τι μελιγενέστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση. Γιατί αποκλείστηκε η Γερμανία. Η Γερμανία δεν αποκλείστηκε. Μας ε, ζητήθηκε να μελετήσουμε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα briefing note, όχι μία λεπτομερής μελέτη, όπως σας είπα και στην αρχή. Συνεπώς ε, διαλέξαμε ε, ένα υποσύνολο των κρατών μελών. Και εξετάσαμε καθένα από τα μοντέλα χωριστά σε συμφωνία με τις ε, υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε ιδιαίτερη μελέτη της περίπτωσης Γερμανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξετάσαμε τη Γερμανία. Συμπεριλήφθη στην ανάλυση που κάναμε, ε, στην, στην, στο briefing note της γενικής ανάλυσης αναφερόμαστε στη Γερμανία. Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν υπάρχει case study, αλλά αυτό συμφωνήθηκε εκ των προτέρων με τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου. Και για να είμαι και τελείω ειλικρινή, το εν μέρη συνδεδεμένο μοντέλο έχει ε, θετικά και αρνητικά ε, σε όλες τις χώρες που το εφαρμόζουν. Συνεπώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, ποια χώρα αναλύουμε υπό την προπόθεση ότι θα αναλύσουμε αυτό το σύστημα. Τώρα, ε, ε, ένας ένας, κυρία Σιρακιάνη καταρχήν. Ρωτήσατε την άποψή μου για τις κάτω χώρες και τη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τις κάτω χώρες, ε, είναι μια χώρα όπου έχουν επέλθει σημαντικέ βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα, στην αξιοπιστία, στην ακρίβεια εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένα δίκτυο με ιδιαιτερότητες και τη δική του δομή. Είναι ένα πυκνό δίκτυο με ε, πολλούς επιβάτες που το χρησιμοποιούν για να πάνε στο χώρο εργασίας τους. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα, σε μερικές περιπτώσεις ναι, παρόλο ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε όλη την Ευρώπη. ορισμένες βέλτιστες πρακτικές θα μπορούσαν να εξαχθούν από όλα τα μοντέλα. Δεν ήταν όμως σκοπός μας να εντοπίσουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές κάθε μοντέλου και να τις ε, ενοποιήσουμε σε ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών. Για τη Γερμανία, από την άλλη μεριά, η Γερμανία έχει ε, σημαντικό άνοιγμα της ε, αγοράς με πολλούς καινούριου παίκτες με πολλές μεγάλες εταιρείε που ήρθαν ε, από τις ΗΠΑ και μπήκαν στην αγορά της Γερμανίας ε, έχουν δοθεί πάνω από 300 άδειε λειτουργία στη Γερμανία αλλά υπάρχουν και πολλά παράπονα ε, προς την Κομισιόν και προς τη Ρυθμιστική Αρχή. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε παράπονα για την DB Energy και θυμάμαι και ε, ότι το θέμα αυτό χρονολογείται εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει σχέση με τις ε, εκπτώσεις ε, για ε, μεγάλες, ε, ε, για μεγάλους πελάτες. Η αλήθεια είναι ότι έχει αναπτυχθεί πολύ η αγορά στη Γερμανία ενώ έχει συρρυκνωθεί στη Γαλλία. Το γερμανικό μοντέλο δίδαξε πολλά πράγματα σε όλους στην Ευρώπη. Θετικά συνήθως, αλλά και ορισμένα λιγότερο θετικά. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι διάβαζα σε μία από τις μελέτες στις οποίες βασιστήκαμε εμείς στην ανάλυση μας, ότι το μοντέλο της Γερμανίας ε, κρισίμευσε ε, μόνο για την οικογένεια της DB. Ε, ευνόησε μόνο την οικογένεια της DB. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει αναλυθεί ε, παρκώς σε προηγούμενες ε, μελέτες. Ο κ. Κούν. Έχετε πέντε λεφτά για όλους τους υπόλοιπους, εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Σε ό,τι αφορά τις ε, χώρες κεντρικής Ευρώπης, η απάντηση είναι ίδια. Συμφωνήσαμε σε μια αρχική επιλογή και αυτήν ακολουθήσαμε. Θα μ' άρεσε και εμένα να έχω συμπεριλάβει πολύ περισσότερες χώρες. Τη Γερμανία, την Ανατολική Ευρώπη, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Το γεγονό είναι ότι είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε χρειάστηκε να διαλέξουμε τις χώρες από τις οποίες είχαμε την περισσότερη, ε, τις περισσότερες πληροφορίες και που αντιπροσώπευαν τα βασικά μοντέλα της Ευρώπης βέβαια. Και τρεμόσα. Γιατί η έκθεση είναι στα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι η ερώτηση δεν αφορούσε εμένα, έτσι. Μα ζήτησαν ναι, η μελέτη να γίνει στα αγγλικά και βέβαια η, ο χρόνος δεν επέτρεπε ε, τη μετάφρασή της προφανώς. Είναι σαφές, δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός ανάμεσα στο μερίδιο αγοράς, στα μερίδια αγοράς και την δομή του μοντέλου. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης μας. Κύριε Κρέιμερ, νομίζω ότι απάντησα σε ορισμένα από τα όσα είπατε. Συμφωνώ πλήρως ε, με τα σχόλια σας για τον, για τον ε, ρυθμιστή. Εμείς ε, αναφέρουμε ότι οι διοικητικές ικανότητες και οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών φορέων είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη τομέα. Ο ρυθμιστικό φορέας θα πρέπει να είναι και επαρκώ επανδρομένο και να έχει επαρκή χρηματοδότηση και να έχει τη σωστή δομή. Δεν είναι βέβαια αρκετό αυτό από μόνο του. Αλλά μία ανοιχτή αγορά με τέτοιο ρυθμιστικό φορέα ε, μπορεί να αναπτυχθεί. Κύριε Ζήλε, πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της μεταφράσης φορτίων. Είναι μια ανοιχτη αγορα με τετοιο ρυθμιστικο φορεα μπορει να αναπτυχθει κυριε ζηλε πω μπορουμε να μειωσουμε το κοστο τη μεταφορα φορτιων ειναι μια καλη ερωτηση αν ο διαχωρισμός μειώνει τις τιμές της μεταφοράς φορτίων. Ε, είναι αμφιλεγόμενο. Στις χώρες που έχουν διαχωρίσει, για παράδειγμα στον Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι τμήμα της μείωσης του κόστους οφείλεται σε αυτό. Θα μπορούσε βέβαια αυτός ο διαχωρισμός ε, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και ίσως αυτό να οδηγήσει σε μείωση κόστους, αλλά δεν υπάρχει άμεσος, άμεση σύνδεση. Σε ό,τι αφορά το πλάτος των ε, γραμμών των τροχιών στις βαλτικές χώρες και στη Φιλανδία, ε, είναι πολύ καλό το σχόλιο. Σε αυτά τα κράτη-μέλη η πρόσβαση είναι, εμποδίζεται και εκεί ίσως υπάρχει μια, ένας τύπος στρέβλος του ανταγωνισμού. Θα πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε από πλευρά διαλειτουργικότητας και όχι σε σχέση με το μοντέλο διαχωρισμένο ή όχι. Αν ο διαχωρισμός οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού, ρωτήσατε εσείς, ε, διευκολύνει τον ανταγωνισμό θα έλεγα εγώ. Δεν είναι ούτε αναγκαίο 100% ούτε επαρκές 100%. Αλλά βλέπουμε ότι εν γέννη, εκεί που γίνεται περισσότερο διαχωρισμός, διαχωρισμός ε, έχουμε και περισσότερο ανταγωνισμό, αλλά δεν έχουμε άμεση σύνδεση και σχέση. Ωραία. Κύριος Ρίκελ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όντως ε, ε, για να σχολιάσω την έκθεση αυτή έχω δύο πράγματα να πω. Αποδεικνύει ότι μετά από 10 χρόνια οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν βοήθησαν καθόλου. Υπάρχει πλήρες χάος όπου όλα τα κράτη είναι, έχουν παραβιάσει τις οδηγίες. Ε, δεν είναι υποχρεωτικά κακή θέληση αλλά στρατηγική που εφάρμοσαν για να παρακάμψουν την οδηγία και χρησιμοποιούν ε, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο σιδηρόδρομος έχει πολύ κακές επιδόσεις. Εμείς εδώ είμαστε υπέρ του σιδηροδρόμου. Θα έπρεπε αντί να ε, υπεραμεινόμαστε ορισμένα πρότυπα να υπεραμεινόμαστε του σιδηροδρόμου και ε, γενικώ ε, είδα ότι υπήρξαν πολλές κατακρίσεις στην έκθεση αυτή. Το δεύτερο που απέδειξε η έκθεση είναι ότι ο όλος ο μηχανισμός λειτουργεί και όχι ένα μέρος μόνο, διότι για την ενέργεια των τηλεπικοινωνιών και άλλων δεν είχαμε θέσει τα ίδια ερωτήματα όπως στους σιδηροδρόμους. Εφαρμόστηκαν συστήματα όπου τα συστήματα εξαρτώνται από, τους, από αυτούς που διεκπεραιώνουν και βλέπετε ότι ο κάθε βάζει το χέρι του και κάνει ό,τι του συμφέρει. Ε, βλέπω ότι ο Μάικλ ασχολήθηκε με τη Γαλλία αλλά η, η ε, Γαλλία, στη Γαλλία έχουμε 50.000 άτομα που ασχολούνται με την υποδομή και στους ε, γερμανικούς συνδεροδρόμους τα ίδια γίνονται οπότε όλοι σε ένα καζάνι βράζουν. Επίσης, αν το είχαμε ξεχάσει μας ε, ε, είπε η μελέτη ότι το σύστημα λειτουργεί καλά. Μας ξαναείπε ότι ο εξυγχρονισμός ε, οδηγεί εις ε, μία πρόοδο η οποία θα πρέπει να ελέγχεται από τους εθνικούς ε, χρήστες και τέλος ότι ο ανταγωνισμός βελτίωσε όχι μόνο τις σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και την ε, ποιότητα και την χρήση του σιδηροδρόμου δηλαδή ο σιδηρόδρομος λειτουργεί πολύ καλύτερα εάν τον διαχειριστεί χειριζόμαστε σωστά και τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στην επόμενη οδηγία. Έχω ακόμη εννέα ομιλητέ και ε, έχουμε τα τελευταία 20 λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν καλύτερα να κάνετε ε, ερωτήσεις για την έκθεση και προσπαθήστε να με βοηθήσετε. Ο κύριος Μπαλτσάιτης. Ευχαριστώ πρόεδρε. συζητούμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και θα ήθελα να συνεχίσω εκφράζοντας τις ιδέες που είχαν ξεκινήσει οι συναδελφοί από την ε, Λετωνία. Λέτε ότι η περίπτωσή μας είναι ενδιαφέρουσα, αλλά το έχουμε δύσκολη κατάσταση, έχουμε διαφορετικό πλάτος γραμμών, διαφορετικό σύστημα διαχείρισης, και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσβαση στις αγορές ε, της Ανατολικής, το Καζακστάν και τις Λιπές. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μια ε, μελέτη για να δούμε κατά πόσον ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο ενσωματωμένο μοντέλο που να αφορά την ζώνη αυτή. Κάποιες δηλαδή χώρες που, που δίνουν αυτές τις προσβάσεις σε ανατολικές αγορές. γιατί εδώ έχουμε και σχέσεις ε, πόρων με τρίτες χώρες και αντίκτυπο αμοιβαίο αντίκτυπο αν θέλετε στα θέματα προϋπολογισμού και κοστολόγησης. Ε, πρόεδρος, να ζητήσω από τους από τα μέλη το εξή. Αν θέλουμε μία μελέτη για τη Φιλανδία, τα βαλτικά κράτη-μέλη κτλ. Έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε. Αυτό δεν ήταν η εντολή που είχε η Steer Davis Cleave. Αν θέλετε να ζητήσετε μια τέτοια έκθεση, ζητήστε την από το συντονιστή σας, ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είχε ανατεθεί αυτή η μελέτη και επειδή δουλέψατε υπό πίεση χρόνου και με συνεχείς αλλαγές όσον αφορά τα διάφορα κράτη και με τον τρόπο που συγκεντρώσατε τα στοιχεία παραδείγματος χάρη εξηγήσατε γιατί δεν έχει ανάλυση της Γερμανίας κατά τη γνώμη μου η εργασία διαδικασία αυτή νομίζω δημιουργεί πιο πολλά ερωτήματα παρά απαντάει και ε, όσον αφορά τις διάφορες αρχές πιστεύω ότι οι ε, αρχές πρέπει να επανδρωθούν με το αναγκαίο προσωπικό όπως άλλοτε επισημαίνεται στη σελίδα 61 αναφέρεστε στην εναρμόνιση και στην εναρμόνιση των κανόνων και των διατάξεων που πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά το κόστος δεν έχετε ε, δώσει ακριβή στοιχεία ε, και πιστεύω ότι η αύξηση του κόστους οφείλεται στην αύξηση των διοικητικών χειρισμών και όσον αφορά την ασφάλεια την αναφέρατε επί, επανειλημμένως σε διάφορες χώρες αλλά γιατί όχι στη Μεγάλη Βρετανία και ουσιαστικά Έχω και άλλα στοιχεία για τα, τα οποία αμφισβητώ πάρα πολύ για τις α, ε, ε, κυβερνητικές αρχές, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία εντυπωσιάζουν και ε, ε, δημιουργούν ερωτηματικά. Ο κύριος Ντιουράν, δύο λεπτά. Η κυρία Ντιουράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα ίσως ε, ε, ε, να ανασκευάσω αυτά που είπε ο κύριος Ρικέ, αν είναι ένα μπάχαλο ή όχι. Διότι υπήρχε μεγάλη ποικιλιομορφία στην Ευρώπη, υπήρχε, υπάρχει ακόμη, το ξέραμε και το ξέρουμε ακόμη. Το να το συγκρίνουμε με τις αεροπορικές μεταφορές ή τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο δεν είναι σωστές παρομοιώσεις. Επίσης δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Δηλαδή είτε υπάρχει ε, ανταγωνισμός και διαχωρισμός ε, μπορεί κανείς να διαχωρίσει τα διάφορα τμήματα της αγοράς. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ο ανταγωνισμός είναι το απόλυτο ιδεώδες αλλά δεν είναι απαραίτητο και αν υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός αλλάζει η στρατηγική, αλλάζει η παιδεία και το κόστος συντονισμού. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε αυτή την, ανασκεύα, ε, ε, στην αναδιατύπωση. Πρέπει να δούμε τι θέλουμε ακριβώς γιατί εάν δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων βλέπουμε ότι δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε κάτι διαφορετικό υποχρεωτικά θα προχωρήσουμε και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ μιλούμε για ένα ε, μέσο το οποίο έχει συγκεκριμένα μερίδια αγοράς ε, ποσοστά δηλαδή και για τους επιβάτες και για την ε, μεταφορτίου. Δεν ξέρω εάν το συμπερασμά μου είναι σωστό, αλλά δεν μας λέτε δεν καταλήγεται σε, σε τελεσίδικο συμπέρασμα σχετικά με αυτήν την αποδηματοποίηση ή unbundling για να συνεννοούμεθα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τελικά δηλαδή όταν μας λέτε ότι αυτή η ο διαχωρισμός αυτών των δύο διαχειρήσεων δεν καθιστά βελτίωση, δεν αντιπροσωπεύει μια βελτίωση ούτε για προς τη μία κατεύθυνση, ούτε προς την άλλη εφόσον έχουμε αύξηση του κόστους κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού, αυτό μπορεί να έχει να σχέση με τις απαιτήσει ε, του ρυθμιστικού φορέα, του συγκεκριμένου κράτους μέλους κτλ. Μας λέτε ότι μπορεί να υπάρχει μια σημαντική αύξηση τιμών. Αρκεί να δούμε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά μαζί μιλάτε και για ανεξαρτησία της λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι διαφορετικό θέμα από το θέμα της αποδεματοποίησης. Μήπως θα έπρεπε να μιλούμε, να έχουμε μια προσέγγιση συνδυαστική και των ελαχίστων απαιτήσεων δηλαδή του κράτους και της ανεξαρτησίας ρυθμιστικής αρχής. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια ε, αρχή σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο ώστε και να εξασφαλίζεται απλώς η ανεξαρτησία σε λειτουργικό επίπεδο. Ε, ο κύριος δύο λεπτά. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. <coughs> Δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση για το θέμα του ανοίγματο της αγοράς αλλά πιστεύω ότι η μελάτη αυτή είναι πολύ καλή και νομίζω ότι ε, ο καθένας βρήκε αυτό που ήθελε όσοι θέλανε unbundling το βρήκανε όσοι θέλανε bundling και, αυτό το, και αυτοί το βρήκαν άρα κάνατε μία μελέτη που ικανοποίησε τους πάντες έχω όμως δύο ερωτήσεις η μία αναφέρεται στη χώρα μου ότι ο Βέλγιο ο ρυθμιστής ούτως ή άλλως πληρώνεται σαν διευθυντής υποδομών και δεν εξετάζεται αν είναι είναι ανεξάρτητος ή όχι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και συνδέεται όμως το γεγονός αυτό με την ερώτηση του συνδέλφου μου Ζορς Μπαχ. Τι εννοείται όταν μιλάτε για ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία είναι νομικός όρος, είναι ουσιαστική ο γεγονός ή μιλάτε και έχετε ελέγξει με την ανεξαρτησία για το εάν υπάρχει και οικονομική ανεξαρτησία γιατί υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που φέρνονται πολύ ανεξάρτητες στα χαρτιά αλλά όταν κοιτάξουμε το κεφάλαιο βλέπουμε ότι υπάρχει σάρα κοιμάρα μέσα. Οπότε δεν είναι μόνο η νομική πτυχή αλλά είναι και η οικονομική πτυχή που πρέπει να ελεγχθούν όταν μιλάμε για ανεξαρτησία. Η ε, κυρία Σελανό ε, για δύο λεπτά. Θα είμαι πολύ σύντομη. να απαντήσω στα όσα είπατε στον κύριο Κούνικ και στον κύριο Κρέμερ. Πιστεύω ότι για να είναι μια μελέτη, πανευρωπαϊκή μελέτη, θα πρέπει να περιλαμβάνονται χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Περιμέναμε πολύ, πολύ καιρό αυτή τη μελέτη και θέλαμε να βγάλουμε πραγματικά αξιόλογα συμπεράσματα. Δυστυχώς αποτύχαμε σε αυτό. Η κυρία Αγιάλα Σέντερς. Συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα στην παρουσίαση των briefing notes. Αλλά είδα τα συμπεράσματα. Η συζήτηση βέβαια έχει εστιαστεί στην διαμάχη μεταξύ των δύο βασικών παρόχων. Ε, είναι κρίμα που δεν έχει συμπεριληφθεί η Γερμανία γιατί αυτό πραγματικά μας δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα. Εγώ δεν θα παραπονεθώ όσες Ω Ισπανίδα που δεν συμπεριληφθήκαμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε διαφορετικό εύρος τροχιών, οπότε στα Πυρηναία ε, υπάρχει σημείο ασυνέχειας είναι σημαντικό να δούμε τα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά το κόστος, αναφέρεται ότι στην περίπτωση του διαχωρισμού το κόστος και η τάση είναι αυξητική. Οπότε η το σημαντικό βέβαια είναι να κοπεί ο ομφάλιος λόρος με τους παραδοσιακούς παρόχους έτσι ώστε να πάμε σε καλύτερες προδιαγραφές ποιότητας αλλά το κόστος ανησυχεί. Πολλές ε, φορές λέτε ότι οφείλεται στην περιπλοκότητα των συμβάσεων. Αλλά ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προτάσεις να επανέλθουμε σε συμβάσεις ολοκληρωμένες. Δηλαδή ε, να επανασυνδεθούν αυτά που παλιότερα είχαν διαχωριστεί. Έχετε στοιχεία για, το, για τους λόγους που, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί για μας ο διαχωρισμός αποτελούσε πάντοτε ε, ένα βασικό συστατικό στοιχείο ενός ευρωπαϊκού μοντέλου. Όχι του γερμανικού ή του ολλανδικού οτιδήποτε. Είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση προς το διαχωρισμό ή μήπως πρέπει να την ξαναδούμε. Θα ήθελα να επανέλθω στα σχόλια στη Γερμανία γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή η παρουσίαση είναι ανόητη διότι έχουμε ε, πάρα πολλούς ε, ιδιωτικούς ε, επιχειρηματίες πλέον της ΔΕΜΠΕ και δεν είχαμε ποτέ απεργίες, κανείς δεν έχει κάνει κάτι ε, για να πάρει πίσω τους πελάτες του, άρα δεν μπορεί το γερμανικό σύστημα να είναι τόσο κακό ως έχει. Να σας δώσω κι εγώ, λέει ο Πρόεδρος, την συνεισφορά μου. Πρέπει να πω στον κύριο Διονόρη ότι θα μπορούσατε να έχετε την καλύτερη έκθεση όλων των εποχών που να έχει υποβληθεί και πάλι εδώ αρκετοί συνάδελφοι θα είχαν βρει ελλείψεις και ελαττώματα και θα σας είχαν επικρίνει. Επομένως αυτές τις επικρίσεις που ακούσατε μην τις παίρνετε και τόσο δηλαδή, πώς να σας πω, μη σας πιάνει η κατάθλιψη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις στην Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τους σιδηροδρόμους τα όρια εδώ που βλέπει κανείς και είναι εμφανή είναι τα εθνικά όρια οι εθνικές ομαδοποίησεις αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση εγώ είχα λάβει και το email από την απάντηση του ΣΥΑ και μετά αμέσως ε, έλαβα την απάντηση και από το SNCF, δηλαδή έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε φορά κάποιος θα διαμαρτύρεται δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση εάν τα μέλη ε, έψαχναν ε, για κάποια κατεύθυνση. Εδώ πέρα το βασικό θέμα είναι αυτή η αποσύζευξη, αυτός ο διαχωρισμός. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ ανέφερε το θέμα ότι το Ηνωμένο Βασιλείο μπορεί να επανέλθει στην σύζευξη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Αλλά το, το συνολικό σύστημα Network Rail δεν ξέρω αν θα επιστρέψει σε τέτοια θέματα επανασύζευξης και αυτό έχει σχέση με εγκατεστημένα συμφέροντα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των γερμανικών σιδηροδρόμων, των γαλλικών σιδηροδρόμων κτλ. Αυτό είναι το βασικό υπόβαθρο, η βασική αιτία. Εγώ έχω την εξή ερώτηση, πάντως. Την ερώτηση που κανείς δεν θέλει να κάνει στην ουσία. Υπό το υφιστάμενο σύστημα που έχουμε στη Γερμανία. Η Γερμανία αντιπροσωπεύει ένα πρόβλημα, είναι πρόβλημα ή μήπω σας δίνει τη δυνατότητα το γεγονός ότι δεν την εξετάσατε τη Γερμανία να μας πείτε κάτι άλλο, να αποφύγετε το θέμα. Και τελικά η γερμανική σιδηρόδρομη για τις υποδομές της λαμβάνει πόρους. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Τι διαφάνεια υπάρχει σε σχέση με αυτό το θέμα. Έχετε 7 λεπτά στη διάθεσή σα, ε, λέει ο Πρόεδρος, και εγώ και εσείς μπορούμε να φύγουμε γρήγορα από εδώ, προτού μας θάψουν με τις <laughs> ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Κοίταξτε, θα ξεκινήσω με το απλούστερο. Θα έπρεπε να έχουμε μελέτη για την ενσωμάτωση των βαλτικών χωρών. Βεβαίω. Αλλά εγώ αυτό θα έλεγα γιατί σύμβουλο είμαι. για τον ε, κύριο Μπαχ. Υπάρχουν αρκετές απαντήσεις που οδηγούν σε περαιτέρω ερωτήσεις σε αυτόν τον τομέα. Προσπαθήσαμε στον λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να δώσουμε όσες απαντήσεις μπορούσαμε, αλλά έχετε δίκιο. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Πράγματι υπήρξαν αυξήσει κόστους. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το είχα αναφέρει και στην παρουσίαση, αυτό δεν σχετίζεται αναγκαστικά με την αποσύζευξη. Είχαμε νέες επενδύσεις, ανανεώσιμα, το οποίο είχε σχέση με έλλειψη επενδύσεως πριν, στην προηγούμενη φάση. Ίσως βέβαια μπορεί κανείς να πει ότι ο διαχωρισμός αποσκοπούσε ακριβώς το να καταστήσει την εικόνα της επιχείρησης ελκυστικότερη ώστε να προσελκύσει επενδύσει, αλλά επ' αυτού δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και απτές αποδείξεις. Πάντως το θέμα της ασφάλεια είναι ευαίσθητο και λεπτό θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ευθύ ε, διασύνδεση μεταξύ αντικτύπου στην ασφάλεια και διαχωρισμού αποσύραξης. Δεν υπάρχει, υπάρχουν ενδείξει για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια άμεση σχέση. Η ε, κυρία Ντιόν δεν νομίζω ότι κανείς δεν θέλει στο πεδίο των σιδηροδρόμων να διαχωρίσει για την αξία του να διαχωρίσει. Καθ' αυτό. Εδώ έχουμε ζητήματα αποτελεσματικότητας, ε, μείωσης του κόστους, αύξηση του ανταγωνισμού και ελπίζουμε βελτιώνοντας τελικά την αγορά για τον τελικό χρήστη, τον επιβάτη ή την εταιρεία που θέλει να μεταφέρει το φορτίο της, το εμπόρευμά της. Δεν είναι η μόνη κατεύθυνση που έχουμε μπροστά μας. Απλώς είναι ένα βήμα που ενδεχομένως να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετική φιλοσοφία και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του ενσωματωμένου σιδηροδρομικού τοπίου. Δεν υπάρχει ίδια φιλοσοφία στην Ευρώπη. Αν δείτε τις τεχνολογικές μόνο διαφορές που ήδη θίξαμε κάπως στην παρουσίαση, καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστεί πολύ καιρό για να τα ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά. Το οποίο είναι θεμελιώδες για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια πιο ανοιχτή αγορά. Για τον κύριο Στέρξ, αυτό το 6% αύξηση στα εμπορεύματα, στις μεταφορές εμπορευμάτων, δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Κάτι ακούμε εκτός μικροφώνου τώρα, μάλλον δεν ακούμε για να είμαστε πιο ακριβείς. Έχετε δίκαιο λέει ο κύριος Διονόρη. Μας τελειώνει και ο χρόνος, λέει ο Πρόεδρος. Είμαστε τόσοι, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε αύξηση κόστους και πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος έλεγχος σε εθνικό επίπεδο, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το έχουμε καλύψει. Για τον κύριο Γκρόσο, μάλλον δεν είναι εδώ ο κύριος Γκρόσο, για τα, της ανεξαρτησίας, την νομική βάση είναι περισσότερο και πάλι θέμα φιλοσοφίας. Η ανεξαρτησία δεν είναι σαν, είναι σαν τον κατακαιρματισμό, δεν το κάνει κανείς αυτό σκοπό. Ε, δίνει κίνητρα επενδύσεων να έρθουν περισσότεροι επενδυτές στην αγορά των σιδηροδρομικών. Αν δεν έχουμε μια επαρκώς ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, δεν υπάρχει η επαρκής ε, βεβαιότητα για να προχωρήσει κανείς σε μια τέτοια επένδυση. Επομένως, επί του θέματος ανεξαρτησίας ε, των πόρων, της χρηματοδοτικής δηλαδή ανεξαρτησίας, δεν το έχουμε δει εξ ολοκλήρου αυτό, αλλά το βασικό είναι να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο και την κατάλληλη φιλοσοφία και προσέγγιση ώστε να προσεγγίσουμε επενδύσεις. Για την κυρία ε, Σεχνάλαβα και το ότι δεν είναι πανευρωπαϊκή μελέτη. Δεν είναι μελέτη καν είναι σημείωμα πληροφόρησης. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε μια ευρύτερη μελέτη στον χρόνο που μας είχε δοθεί. Δυστυχώς. Για τον κύριο Κόχ και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά ή τις διακρίσεις αντίστροφα. Εδώ μιλούσαμε για παραβάσεις, όχι καταγγελίες αναγκαστικά. Έχουμε αρκετές διαμαρτυρίες και καταγγελίες στη Γερμανία από ανθρώπους που θέλουν πρόσβαση. Και εδώ επανέρχομαι στην βεβαιότητα. Δυνητικά θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερα τέτοια περιστατικά, γιατί δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας βεβαιότητας στον κλάδο. Κάτι πάλι ακούγεται εκτός μικροφώνου από τον κύριο Κράμα. Τελικά η μη χρησιμοποίηση της Γερμανίας είναι πρόβλημα ή δικαιολογία λέει ο πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα, λέει ο κύριος Διονόρη. Είναι θέμα προτύπων, μοντέλων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την μελέτη μας, για την εξέτασή μας. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη εξέλιξη σε όλες τις αγορές. Όλες οι αγορές αλλάζουν και εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν υποτένει αυτοί, αυτή, τα πρότυπα που κυριαρχούν στα διάφορα κράτη-μέλη, τις θετικές και αντικές πτυχές τους και θα μείνω σε αυτά, Πρόεδρε. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Ντιονόρη. Πράγματι, όπως βλέπετε, είναι κάτι που ενδιαφέρει έντονα τα μέλη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Οι τροπολογίες ή μάλλον το χρονοδιάγραμμα έχουμε το σχέδιο έκθεσης για τις 24 Μαΐου, την εξέταση των τροπολογιών για τις 20 Ιουνίου, ψήφιση 20 Ιουλίου στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Και νομίζω 30 Μαΐου ήταν η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και χθε το βράδυ, το λέω στον κύριο Τριμόσα, επιβεβαίωσαν το χρονοδιάγραμμα και οι συντονιστέ, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Δεν έχω άλλα στην ημισία διάταξη, εκτός από το να σας πω ότι ε, η επόμενη συνάντηση θα είναι Βρυξέλλες, 23 Μαΐου, στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστεί ευγενικά ο πρόεδρος ε, Διερμηνής, ευχαριστούμε και εμείς. Λήξη την συνεδρίαση.